Dear colleagues, ladies and gentlemen. Ξεκινάμε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες καθώς και κύριοι. I will start Θέλω να σας κάνω ορισμένε ε, ανακοινώσεις πρώτα. Πρώτα απ' όλα. Η Επιτροπή μας θα συνεδριάσει στο Λουξεμβούργο στις 3 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεκτικό ε, συνέδριο. Θα τα κανονίσει αυτά η γραμματεία και θα σας δώσει πληροφορίες εν καιρό. Έχω να ανακοινώσω επίσης τους εξή διορισμούς. Ο κύριος Ζιδιεύκα από το ΕΛΚ θα είναι ο εισηγητής για την άρση της κοινοβουλευτικής ε, ασυλίας του Ιβαν Γιάκοφτσιτς της Αλδε, Ο Ζω Καβαντά από την Αλδε αρμόδιος συντονιστής για την ομάδα εργασίας για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μεταρρύθμιση του copyright, η Heidi Hautala από τους Πράσινους θα είναι μόνιμη συγγήτρια για τα θέματα διοικητικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μέλος των σοσιαλιστών θα είναι εισηγητής για το πρόγραμμα REFIT, Regulatory Fitness κτλ για τα, τις μελλοντικές προοπτικές του Ριφίτ. Επομένως, εγώ η ταπεινότης μου θα είμαι εισηγητής για την ε, νέα συνένεση σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ροζιέρα από τους σοσιαλιστές θα είναι η κυρία Ροζιέρα, συγγνώμη, θα είναι εισηγήτρια για την παράταση του καθεστώτος γεωγραφικής προέλευσης για μη γεωργικά προϊόντα. Η Γιούλια Ρέντα από τους Πράσινους εισηγήτρια για την εφαρμογή της οδηγίας 2001 κάθετος 29 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του copyright και συναφών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Ένα μέλος της ECR, της Συνδετική και Μεταρρυθμιστικής Ομάδας, θα είναι αρμόδιος για τις αιτήσει εκθέσεις 2012-2013 σε σχέση με την επικορικότητα και την αναλογικότητα. Από την ΚΟΕΘ θα είναι κάποιος εισηγητής για την 30η και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έτη 2012 αλλά και 2013 συμπεριλαμβάνοντας τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητος σε σχέση με την εφαρμογή της πρωτογενούς νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς θα προσκληθεί σε μια ε, συνεδρίαση στο μέλλον της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή μας επίσης θα συνδεθεί μαζί με την ακρόαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μια ακρόαση που θα γίνει στην αρχή του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τεχνολογίες τον αντίκτυπο της ε, ψηφιακής παρακολούθησης και των συστημάτων διείσδησης. Και προσκαλείστε να είσαστε παρόντες στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ετήσιας ε, συνδιάσκεψης των διευθυντών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα λάβει χώρα στις 11 Δεκεμβρίου για θέματα εκπαίδευσης και αυτό υποστηρίζεται από τις Επιτροπές ε, Νομικών Θεμάτων και ΛΥΜΠΕ. Θα στείλουμε επίσης μια επίσημη επιστολή στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων για να υπάρξει μια επίσημη ερμηνεία των, της λέξης σκρούτινη όπως χρησιμοποιείται στο παράτημα 1α του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά είναι οι ανακοινώσεις μου λοιπόν. Περνάμε τώρα στο σημείο 41 το οποίο αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη διαδικασία αφαιρεγγιότητος και με μεγάλη χαρά θα δώσω εδώ το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Ζηλιέφκα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, χτες έγινε συνεδρίαση, ένας τριμερής διάλογος που ολοκλήρωσε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν τον κανονισμό για την φερεγγιότητα. Να υπενθυμίσω εν συντομία συνάδελφοι ότι οι συζητήσεις επί του κανονισμού ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της πρώτερης θητείας. Ο κύριος Καλ Χάινε Λένε ήταν ο εισηγητής. Είχα το προνόμιο να συνεχίσω το δικό του έργο το κείμενο που ετοίμασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα δύο κείμενα ήταν πολύ κοντά σε αρκετά θέματα, όμως υπήρχαν και αποκλίνουσες απόψεις επί άλλων σημείων και γι' αυτό έπρεπε να προβούμε στη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης και έπρεπε να γίνουν διάφορες διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν χτες. Δύο στοιχεία ή ε, απετέλεσαν αντικείμενο των προσπαθειών μας. Θέλαμε το Συμβούλιο να αλλάξει τη θέση του, να λάβει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά. Το πρώτο σημείο ήταν το άρθρο 3 που αφορούσε τη δικαιοδοσία. Πάντα προσπαθούσαμε αυτή την πτυχή να τη λαμβάνουμε υπόψη. Πάντα είχαμε στόχο τον περιορισμό των κινήτρων ούτως ώστε κάποιος να ε, προσπαθήσει να διαλέξει ε, κάποια δικαιοδοσία όπου θα μπορούσε να ευνοηθεί ένα μέρος των αντιδίκων, μια πλευρά. Λόγω της νομοθεσίας της ε, χώρας ή λόγω των αρμοδίων φορέων. Δεν θέλαμε να υπάρχει, να γίνεται το λεγόμενο foreign shopping σε αυτό το τομέα, το τελικό κείμενο που απέρευσε από τις διαπραγματεύσεις ικανοποιεί τις προτιμήσεις μας και η αιτιολογική σκέψη, η 12 ε, που αφορά τα ίδια ζητήματα, άλλαξε ούτω ώστε να συνάδει με το άρθρο 3. Το δεύτερο θέμα που ήταν εστία των προσπαθειών μας ήταν η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, μια πρόταση του κυρίου Κονφεράτη, όπου προσπαθούσαμε να δώσουμε ειδική προστασία στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια των ε, διαδικασιών ε, για την αφαιρεγκαιότητα. Αυτή η αναφορά έλειπε από το αρχικό κείμενο, αλλά όλοι συμφωνούσαμε, συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται. Μετά από πολύ δυσχερείς διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, κατορθώσαμε χτες να υιοθετηθεί αυτή η θέση μπορούμε να πούμε τώρα ότι σαν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο έχει πετύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους κοιόδης εισηγητές, τον κύριο Κομφεράτη όλος ιδιαίτερος και τον κύριο Μαρίνιο Πίντο που συμμετείχαν και οι δύο στις προπαρασκευαστικές εργασίες και στις ε, ε, συνομιλίες του τριμερούς διαλόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας στο έργο μας και ακολουθήθηκε πολύ θετική προσέγγιση από πλευράς Ιταλικής Προεδρίας. Η Ιταλική Προεδρία κατάφερε να πείσει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρόλο που δεν ήταν εύκολο το έργο. Μετά την ε, περάτωση του τριμερούς διαλόγου χτες έχουμε την εξής κατάσταση. Περιμένουμε το Συμβούλιο να μας δώσει ένα ενοποιημένο κείμενο μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, το αργότερο. Ούτως ώστε στις 2 Ιανουαρίου, κατά την επόμενη σύνοδο της Επιτροπής μας, θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε την τελική εκδοχή του κειμένου. Να το εγκρίνουμε στην Επιτροπή. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει το κείμενο το Δεκέμβριο και αυτό σημαίνει ότι θα υποβληθεί το κείμενο στην Ολομέλη αρχές του επομένου έτους για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ όλους και χαίρομαι όλους ιδιαιτέρως που αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα κατέληξε θετικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τις θετικές αυτές πληροφορίες. Στο ίδιο σημείο να δώσω το λόγο στον Μπρούνο Πάολη που εκπροσωπεί την Ιταλική Προεδρία. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και την ευκαιρία και εγώ να συνεχίσω αυτά που είπε και ο Σβιέσκα. Είμαι ικανοποιημένος που μπορώ να ανακοινώσω ότι πράγματι πετύχαμε μια συμφωνία. Δεν ήταν κάτι δεδομένο, αυτό μπορούμε να το προσθέσουμε. Όπως είπε ο κ. Βιέσκα, πρόκειται περί κανονισμού σημαντικότατου για το οικονομικό μέλλον των ε, επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως στιγμές κατά τις οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και αυτός ο κανονισμός έχει ένα ισχυρό σημείο, σημαντικότατο, ε, δηλαδή αντιστρέφει την όλη προπτική την οπτική γωνία από την οποία εξετάζουμε τη φερεγγιότητα των επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες δεν πηγαίνουν προς τη ρευστοποίηση πλέον, αλλά θέλουμε να δώσουμε ε, δεύτερη, δεύτερη ευκαιρία στον επιχειρηματία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό όσον αφορά τον κανονισμό. Θα ήθελα να πω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, ήταν δύσκολες γιατί ήταν πολύ περίπλοκο το κείμενο. Εντός του κειμένου, άλλων επί του κειμένου έγιναν διαπραγματεύσεις, ήταν πολλές οι ώρες, μέρες και νύχτες που συνεχίστηκαν και που γινόταν οι ε, διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες δεν ήταν οι πλευρές έτοιμες ακόμα. Το αποτέλεσμα τριμερούς διαλόγου δείχνει ότι όταν οι δύο συνομοθέτες δρούν ε, με ρεαλιστικότητα, με ειλικρίνεια και καταβάλουν προσπάθειες μπορούν να γραφτούν και ωραίες όμορφες σελίδες της ιστορίας της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Όπως είπε και ο κύριος Βέσκα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υποβάλει αιτήματα το Συμβούλιο επί μακρόν συζήτησε τα αιτήματα αυτά. Πρέπει να πω ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Δεν ήταν εύκολο να πείσουμε το Συμβούλιο να δεχτεί κάποια αιτήματα που όμως όπως έλεγα λόγω επευθυνότητας που διάκρινε τη συνεργασία τη διαθεσμική τελικά έγιναν δεκτές οι προτάσεις και το Συμβούλιο δέχτηκε να τροποποιήσει το κείμενο για να μπορέσει να λάβει υπόψη τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσία το Κοινοβούλιο, τον συγητή, τους σκιώδεις συγητές για την ευαισθησία που επέδειξαν και για τη διαθεσιμότητά τους. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ επαγγελματική υποστήριξη που μας παρήχε και όπως έλεγε και ο κύριος Βέσκα, ε, τώρα είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 4 Δεκεμβρίου να καταλήξει σε θέση. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ με την αισιόδοξη νότα των λόγων του κυρίου Βουλευτού για ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο επετεύχθη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. I think... Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σιέφκα και την Ιταλική Προεδρία για τα θετικά αυτά νέα. Και τώρα μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο υπαριθμό 11, ανταλλαγή απόψεων για την εταιρική διακυβέρνηση. Και εδώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοφεράτη. Μια στιγμή μονάχα λέει ο κ. Μαρτίνιου Πίντσου. Στο σημείο 11 ή δυνατόν θα ήθελα να διαβάσω μια δήλωση της κυρίας και κυρίας Βίξτρομ η δυνατον θα ηθελα να διαβασω μια δηλωση της κυριας και κυρία βιξτρομ η οποια μου ζήτησε να το πράξω αυτό υπό μορφή εισαγωγή στο σημείο αυτό. Ας δώσουμε όμως πρώτα στον εισηγητή το λόγο και μετά μπορείτε να διαβάσετε αυτή τη δήλωση κύριος Κοφεράτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλάμε για ένα θέμα που συζήτησε η Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων, αλλά είναι πιο ευρύ το θέμα που αφορά τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Να πω στους συναδέλφους ότι πρόκειται περί του ζητήματος κυρίως για τη μελλοντική προπτική του οικονομικού συστήματος και για τα αγαθά και έτσι υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πιστεύω ότι ακολουθήθηκε ε, μία λογική ε, ε, που δεν εξέτασε πολύ λεπτομέρειε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των επιχειρήσεων και όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, μετόχων. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα παλιά όρια. Είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς την επιχείρηση ε, και όλους τους εμπλεκόμενους σε μια επιχείρηση και όχι τους μετόχους μόνο θα πρέπει όσον αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβουμε υπόψη. Που θα πρέπει η επιχείρηση να προβάλλει τον εαυτό της στο μέλλον. Που εργάζεται όχι μόνο να έχει βραχυπρόθεσμα ε, κέρδη και να, τα, να μοιράζει το μέρισμα στους μετόχους, αλλά πρέπει να ακολουθείτε ε, να λαμβάνεται υπόψη και το δόγμα της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης. Θα παράγεται πλούτος και έσοδα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες του κράτους, της περιφέρειας ε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στα συμφέροντα όλης της Ένωσης. Λοιπόν, ξεκινώντα από όλου του εμπλεκόμενου και από του εργαζομένου που εργάζονται στην επιχείρηση και σε αυτού πρέπει να δοθεί επαρκή ε, προσοχή. Και όσον αφορά τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλου, θα πρέπει να, καλύπτονται και αυτοί και στη δομή της επιχείρησης, αυτούς που συμμετέχουν στη δομή της επιχείρησης. Σε κάποιες έχουν, υπάρχουν συμβούλια εποπτείας στην επιχείρηση, στα διοικητικά συμβούλια έχουν παρουσία, υπάρχει παρουσία των εργαζομένων, οργανωμένη των εργαζομένων σε αυτούς τους φορείς και ελπίζω αυτό να γίνει γενική τάση του ευρωπαϊκού μοντέλου της διοίκησης που θέλουμε να θεσπίσουμε για το μέλλον. Λοιπόν, υπάρχουν όρια στην πρώτη προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Ελπίζω να ξεπεραστούν τα όρια σύντομα, να γίνει ευρύτερο το πλαίσιο. Η πρόταση Ευρωπαϊκής επιτροπή δεν περιέχει όμως κάποια χρήσιμα στοιχεία, σημαντικά στοιχεία, παρόλο που προσανατολίζονται αποκλειστικά προς τους μετόχους. Ποια είναι τα χρήσιμα στοιχεία. Μεγαλύτερη διαφάνεια προτείνεται όσον αφορά τη συμπεριφορά των μετόχων, το πώς λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και θα πρέπει να οθούν κίνητρα ούτως ώστε οι επιλογές των επιχειρήσεων και των μετόχων να κατευθύνονται προς μία μεσοπρόθεσμη ε, προσέγγιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζεται και αρνητικά από ένα σύστημα. Διάφορες συμπεριφορές οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά η όλη συμπεριφορά ε, αφορούσε τα σύντομα κέρδη. Μερίσματα για τους μετόχους, για αμοιβέ για τα ανώτατα στελέχη. Βραχυπρόθεσμα ήθελα να πετύχουν ισχυρή οικονομική θέση, χωρίς να κάνουν μακροπρόθεσμη προβολή, ακολουθώντας κριτήρια σωστά. Όπως ε, οι όροι για την κοινωνική ευθύνη που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 90. Αυτές οι αρχές ακολουθούν, αλλά είναι ξεπερασμένες πια πρέπει να εξετάσουμε τις θετικές πτυχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά να προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε την πρόταση με τα αποτελέσματα των συζητήσεων και των προτάσεων των συναδέλφων. Ξεκινώντας από τι απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Η αφετηρία είναι μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Και θα πρέπει να δούμε και ποια προσέγγιση ακολουθούν οι μέτοχοι που επενδύουν επιχειρήσεις. Παίζουν και θεσμικό ρόλο οι μέτοχοι. Δεν είναι, οι μέτοχοι. Δεν είναι απλώς ιδιώτες. Θα πρέπει να βελτιωθεί δυνατότητα ψηφοφορίας από πλευράς των μετόχων. και εκτός των ιστορικών ορίων που έχουν τεθεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μετόχων και των διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης. Έτσι διευκολύνει τη διαβίβαση των πληροφοριών που καθορίζουν και τις συμπεριφορές. Να υπάρχει σωστή μεταβίβαση των πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το μήκος αλυσίδας της διοικητικής. να μην κινούνται, ε, να λαμβάνονται υπόψη και άλλες τυχές στρατηγικές αποφάσεις που παίρνουν οι επιχειρήσεις. Κάτι που δεν γίνεται τώρα. Είναι ένα στοιχείο αδυναμίας αυτό που δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση και μπορεί να ξεπεραστεί αυτό μέσω ενός συστήματος διαβίβασης πληροφοριών, συνεχούς διαβίβασης πληροφοριών που να δείχνουν ποια είναι η πορεία που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις. Πρέπει να αναπτυχθούν και μηχανισμές που αποφεύγουν τις καταχρήσεις ε, με τις σχέσεις με τους διάφορους συσχετιζόμενους φορείς. Καμιά φορά αλλάζουν σχήμα οι εταιρείε και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στους μετόχους. αλλάζουν κατεύθυνση της επιχείρησης χωρίς να λαμβάνεται μια επίσημη απόφαση από όλους, χωρίς να δίδεται μια ιδέα του επιδιωκόμενου στόχου με συμμετοχή ε, όλων των εμπλεκομένων. Οι μορφές ερινές ελέγχου δεν είναι αποτελεσματικές. Πρέπει να βελτιωθούν τα συστήματα ελέγχου. Και όταν μιλάμε για διαφάνεια, εν γέννη, θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα να γνωρίζονται και διάφορες αλλαγές που γίνονται όταν αυτές υλοποιούνται σε επιχειρήσεις. Χρειάζεται αποτελεσματικό μηχανισμός α, να έχουν λόγο οι μέτοχοι και όσον αφορά και τις αμοιβέ που παίρνουν τα διοικητικά στελέχη. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, δίνει κίνητρα στους, ε, στα διοικητικά στελέχη, αλλά επηρεάζει και τη ζωή μιας επιχείρησης. Πρέπει να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της αμοιβή και των επιδόσεων. Πολύ συχνά δεν γίνεται αυτό. Η σχέση λοιπόν ε, επιδόσεων με, της επιχείρησης με αμοιβέ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αμοιβή των εργαζομένων. όσον αφορά τα ηγετικά στελέχη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που περνάνε φοβερή κρίση όπου καταβάλλονται πολύ ψηλές αμοιβέ στα διοικητικά στελέχη με αυξανόμενη διαφορά. Πάει άσχημα η επιχείρηση και αμείβονται όλο και περισσότερο με αμοιβέ έκτακτε τα διοικητικά στελέχη χωρίς λόγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να το εξετάσουμε για να εισάγουμε ε, σωστά ε, στοιχεία και να μην συνεχιστεί αυτή η πρακτική που ήταν πολύ επιζήμια για πάρα πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα σταθώ εδώ για την ώρα. Ήθελα να φέρω κάποια σημεία που θεωρώ ότι έχουν προτεραιότητα. Μετά θα έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε άλλες συζητήσεις που θα γίνουν, να τα εξετάσουμε αυτά. Βασίζομαι πολύ στους συναδέλφους ξεκινώντας από τους Σκιώδης να συμβάλλω στη συζήτηση, να υπενθυμίσω εντάχει το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μια κρόαση για την οδηγία θα, στις 2 Δεκεμβρίου, παρουσίαση του σχεδίου κειμένου, σχεδίου εκθέσεως στο δεύτερο εξάμεινο του Ιανουαρίου και η προθεσμία της τροπολογίας είναι αρχές Φεβρουαρίου. Μετά θα κάνουμε τα υπόλοιπα και ενδεχομένως θα εγκριθεί το κείμενο τέλος Μαρτίου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να κάνουμε προσεκτική δουλειά, όπως πάντα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και αρκετά γρήγορα. Η ταχύτητα δεν πρέπει να αποκλείει την εμβάθυνση και την προσοχή των θεμάτων που θα θεωρήσετε ότι είναι τα πιο σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο λέω στους συναδέλφους και κυρίως τους κοιόδης ότι πέρα από τον χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει για τις συζητήσεις είμαι στη διάθεσή σας για άμεσες συζητήσεις μαζί τους, διμερείς επαφές για όλα τα θέματα που θα ήθελαν να τα εξετάσουν εις βάθος κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο κ. Μαρίνιου Πίντου ο οποίο επιθυμεί να, δηλώσει, να διαβάσει δήλωση της κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Κοφεράτη. Μου ζήτησε η κυρία Βίξτρομ να εκφράσω την ε, λύπη της για το γεγονός ότι κολλείεται και δεν μπορεί να είναι παρούσα, αλλά αυτή τη στιγμή προεδρεύει της Επιτροπής Αναφορών. Ήθελε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον κύριο Κοφεράτη και με άλλους συναδέλφους σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα. Η ομάδα των φιλελευθέρων θέλει να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση και αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την ενίσχυση των οικονομιών <clears throat> ιδίως μέσα στην οικονομική κρίση που, διερχόμαστε. Αυτά ήθελε να πει η κυρία Σεσίλια Βίξτρομ. Σας ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Ο κύριος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Απλώς θα ήθελα από τη μία πλευρά να αποτίσω φόρο τιμή στο έργο του κυρίου Κοφεράτη και για τον σαφέστατο τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιάσει τα διακυβευόμενα στο θέμα αυτό και θέλω να το διαβεβαιώσω για την πλήρη υποστήριξή μας για το θέμα αυτό και το γεγονός ότι θα τον υποστηρίξουμε πλήρως Θέλω να σταθώ τώρα σε ένα σημείο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή σε σχέση με το εταιρικό δίκαιο στην Ευρώπη, γιατί περνάμε από ένα κόσμο του επιχειρήν σε ένα κόσμο όπου επικρατεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Και αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί ιστορικά ο επιχειρηματίας είχε μια μακροπρόθεσμη, μια μακροχρόνια αντιμετώπιση. Ήθελε να δημιουργήσει πλούτο για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για τους εργαζομένους του, για τη χώρα του, που θα είχε χρονική συνέχεια. Αυτή η λογική τώρα αλλάζει, γιατί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδιαφέρονται μόνο για την απόδοση των επενδύσεων και αυτό είναι κάτι το βραχυχρόνιο. <clears throat> Εδώ για τη διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων οικονομικέ συγκρούσει συμφερόντων. Ο καθένα έχει το δικό του ρόλο μέσα σε αυτέ τι συγκρούσει. Απλώ θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε μια νέα ισορροπία μεταξύ των εμπλεκομένων, των εργαζομένων, των μικρομετόχων και τονίζω ότι το ρόλο των ε, ε, εργαζομένων. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια επιχείρηση ενάντια στους εργαζομένους που είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν την προσθέμενη αξία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και είναι από τα προβλήματα του 21ου αιώνα πώς θα εξασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα σε μια βραχυπρόθεσμη θεώρηση και στην απαραίτητη μακρό, μακρόπνοη αντιμετώπιση και αυτό δεν είναι μονάχα ένα οικονομικό θέμα αλλά και ένα πολιτικό θέμα. Ζιεύκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Λαϊκού κόμματο, ως εισηγητής έχει αναλάβει ο κύριος Τόντ, αλλά δυστυχώς είναι απόν σήμερα και έτσι μου ζήτησε να μεταφέρω τις ευχαριστίες του στον κύριο Κοφεράτη, τον εισηγητή, καθώς επίσης να διαβεβαιώσω τον κύριο Κοφεράτη ότι η πολιτική μας ομάδα θα τον υποστηρίξει. Θα υποστηρίξει τι προσπάθειές του για την επίτευξη ενός ισορροπημένου αποτελέσματος, διότι ο στόχος που έχουμε ενώπιόν μας είναι να ενισχύσουμε τους δεσμούς, την διασύνδεση δηλαδή, μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων των ε, ηθινόντων των επιχειρήσεων για να εξασφαλιστεί η υγεία των επιχειρήσεων. Έδειξε και η κρίση πόσο απαραίτητο είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ ότι οι αυξανόμενες αμοιβέ, τα μπόνους των μελών των διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, ενώ η ίδια η επιχείρηση πάει από το κακό στο χειρότερο, είναι απολύτως απαράδεκτα. Ο κύριος Τόντ τονίζει επίσης ότι οι στόχοι που επιθυμούμε να επιτύχουμε με την λογοδηγία... μπορούν να εφαρμοστούν και με την εφαρμογή της αρχής Save and Play. Μας ζητεί επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς προχωρούμε στις αλλαγές αυτές, διότι στην αρχική πρόταση περιλαμβάνονται στοιχεία που ίσως να έχουν αρνητική επίπτωση στην λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. και στην μακροπρόθεσμη δημιουργικότητά τους και έτσι να μειωθεί η ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά. Η διάταξη που επιτρέπει στην μειοψηφία των μετόχων να έχουν μεγαλύτερη επιρροή σε συναλλαγές με άλλες συγγενείς επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπλοκή των μειοψηφούντων αυτών μετόχων στην διεύθυνση της επιχειρήσεως. Ο κύριος Τότ, λοιπόν, πάντοτε διαστόματός μου, τονίζει ότι σε ορισμένες χώρες μέλη ισχύουν ήδη κάποια, κάποιες νομικές προβλέψεις που επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την διασύνδεση για την οποία μιλούσα προηγουμένως. Και επομένως και έναν ένα επαρκές επίπεδο ελέγχου. Το ίδιο και η οδηγία για τις προφορίες που δίνονται στις μετόχους για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι σε συνεργασία με τον εισηγητή και σε συνεργασία με τους υπολείπους συναδέλφους της Επιτροπής μας θα καταστεί δυνατό να συντάξουμε πρόταση που να διορθώνει τα εφιστάμενα σφάλματα και να οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο κ. Χόιερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σιγητά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον που δείχνετε και τον χρόνο που αφιερώνετε στο σημαντικό αυτό νομοθέτημα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2014. Πριν προχωρήσω στην πρόταση, είναι χρήσιμο να σας δείξω μερικές διαφάνειες για το πλαίσιο. Και όπως είπαν ορισμένα μέλη σας, τα πράγματα δεν έχουν προκύψει από το πουθενά. Είναι νομοθέτημα το οποίο ξεκίνησε από την οικονομική κρίση. Μετά από δύο μεγάλες διαβουλεύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αδυναμίες των ε, εταιριών, των μεγάλων επιχειρήσεων, που οδήγησαν επίσης και αυτές με την σειρά τους στην κρίση. Και η νομοθεσία για το big banking που εγκρίθηκε πέρσι προβλέπουν επίσης και ορισμένες ε, διατάξεις για τις μεταρρυθμίσεις της corporate governance. Όπως γνωρίζετε, φέτος εξέδωσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, το, για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση τη οικονομία τα είπαν αυτά προηγουμένω ορισμένοι δικοί σας, και ορισμένες συγκεκριμένες δράσει Από αυτές κάποιες ήταν και η αναθεώρηση για την εμπλοκή των μετόχων. Είναι σαφές επίσης ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον της κοινωνίας για την οδηγία αυτή, διότι υπάρχουν και άμεσα και έμεσα στοιχεία όπως είπε και ο εισηγητής σας, διότι μεγάλος αριθμός μετόχων ενδιαφέρονται και αφορώνται κιόλας από τις αλλαγές αυτές. Η ανακοίνωση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του Μαρτίου φέτος έχει ως στόχο να απελευθερώσει περισσότερες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να μειώσει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις τράπεζες και να ενισχύσει τις κεφαλαιοαγορές μας και τις ε, αγορές μετοχών. Δεν θα εξηγήσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εκεί εντάσσεται και αυτή η λεγόμενη corporate governance, η διοίκηση επιχειρήσεων. Έτσι εδώ τα κυριότερα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει, από τις διαβουλεύσεις που κάναμε δηλαδή με τους ενδιαφερομένους, αναφέρονται στην διαφάνεια που βλέπετε. Και το πρώτο, βεβαίως κρούω ανοιχτές θύρες, διότι αυτά τα έχουν πει και άλλοι, ήταν ε, ανεπαρκής η μακροπρόθεσμη κυριότητα των επιχειρήσεων, ownership δηλαδή, και εμπλοκή των μετόχων. Βεβαίως όλοι οι μέτοχοι είναι σημαντικοί, ιδίως όμως οι μεγάλοι μέτοχοι, όπως τα μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία, ε, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Εγώ που έχω ας πούμε 100 μετοχές της ΣΕΛ, είμαι σημαντικός κι εγώ, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική βαρύτητα, τότε η μεγάλη αυτή μέτοχη θεσμική μέτοχη, δηλαδή, είναι πιο σημαντική. Τώρα, είδαμε ότι συχνά είναι τέτοιοι τα συνταξιωτικά ταμεία που δεν εξετάζουν συχνά τις μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες δυνατότητες των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύουν και δεν έχουν και μια μακροπρόθεσμη σχέση με τις επιχειρήσεις αυτές που μπορεί να οδηγήσει σε πιο θετικά αποτελέσματα. Και έτσι δεν στοχεύουν επαρκώς τέτοιου είδους μέτοχοι σε ένα διάλογο και σε μια συνεργασία με την επιχείρηση και επιχείρηση με τους μετόχους. Άλλο σημαντικό στην οικονομική κρίση ήταν ότι οι θεσμικοί επενδυτές και οι asset manager δεν ελέγχουν αρκετά τους ε, διοικητές των τραπεζών, οι οποίοι τελικά οδηγήθηκαν σε ανάληψη σημαντικών κινδύνων, που όπως ξέρουμε οδήγησαν σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε βέβαια και ορισμένα νούμερα στην μελέτη αντικτύπου μας. Πάντως, η απόδοση των χαρτοφυλακίων είναι σημαντική, της τάξης του 72%, δηλαδή 72% των μετοχών που διαθέτουν οι asset manager πολλούνται κάθε χρόνο και αγοράζονται νέες. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν πολύ το τι κάνει η επιχείρηση. Άλλο Άλλη ανησυχία είναι ο ρόλος των συμβούλων, επιχειρήσεων συμβούλων που είναι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν συμβουλές στους μετόχους τι στάση να τηρήσουν στις ε, συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες. Τίθεται και θέματα μεθοδολογίας, τι γίνεται επίσης σε περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων των επιχειρήσεων αυτών. Όπως λέχθηκε και πριν, υπάρχουν και άλλες μεγάλες ανησυχίες για, την, ε, για τις αμοιβέ των ανώτατων στελεχών. Πρώτον, εδώ δεν υπάρχει επαρκή διαφάνεια. Δεν ήταν σαφείς ούτε συγκρίσιμες το τι δίνεται δηλαδή ως αμοιβή στους ε, top managers. Και επίσης η δυνατότητα από πλευρά μετόχων να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις. Να έχουν δηλαδή εποπτεία επί των αμοιβών και να πούν όχι δεν ψηφίσαμε εμείς τέτοιες αμοιβέ. Καμιά φορά δεν είναι επαρκής και καμιά φορά είναι και ανύπαρκτη η δυνατότητα αυτή από πλευρά μετόχων. Επομένως δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ απόδοσης και αμοιβή. Άλλα που μας ανησυχούν είναι οι ε, συναλλαγές με συγγενεί επιχειρήσεις. Πάλι εκεί δεν, υπάρχουν, ε, επαρκή, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος των ε, μετόχων. Τέλος, ανησυχίε σχετικά μέσα στον ε, στην αλυσίδα επαφών μεταξύ και επιχειρήσεως και των μετόχων. Δεν γνωρίζουν οι επιχειρήσεις συχνά ποιοι ακριβώς είναι οι μέτοχοι. Το ίδιο δύσκολο είναι για τους μετόχους να ασκήσουν τα δικαιώματά των. Εγώ δίνω πάντα το ίδιο παράδειγμα. Εάν έχω στην κατοχή μου μετοχές σε μια επιχείρηση, ας πούμε στη Γαλλία, και θέλω να ψηφίσω με αυτές τις λίγες μετοχές που έχω, πρέπει να πάω στην τράπεζά μου, η τράπεζα στέλνει ένα τέλεφαξ, τέλεφαξ ναι, σε άλλη τράπεζα και ούτω καθεξής. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ανάγκη να ομαλοποιηθεί η αλυσίδα αυτή επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων, των μετόχων και, το, των επενδυτικών επιχειρήσεων. Οι συγμένε επιχειρήσει επίση αντιμετωπίζουν βεβαίω πολύ σημαντικέ βραχυπρόθεσμε πιέσει. και όταν κανεί αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμε πιέσει, την είναι αγνοεί το μακροπρόθεσμο. Επομένω δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική, στη στρατηγική σου. Επίσης, οι μέτοχοι έχουν δυσκολίες, όπως είπα πριν, να ασκήσουν τα δικαιώματά των και αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει αρκετή εμπλοκή μεταξύ μετόχων και επιχειρήσεων, χάνεται ένα σημαντικό δυναμικό για ολόκληρη την κοινωνία. Τώρα, η πρόταση, ε, συντομεύω, Πρόεδρε, τα βασικά στοιχεία της προτάσεως. Πρώτο, ταυτοποίηση των μετόχων. Σημαντική. Διότι Υπάρχουν τόσοι πολλοί ενδιάμεσοι στην αλυσίδα αυτή που είναι μακρότατη ανάμεσα στην επιχείρηση και στον μέτοχο. Και αυτό περιπλέκει τα πράγματα, προφανώς. Προτείνουμε λοιπόν η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας που είναι η τράπεζά της να εντοπίσει, να ταυτοποιήσει τους μετόχους. Έχουμε και κάποιες τεχνικές ιδέες βέβαια για το πώς να απελευθερώσουμε αυτή τη ροή πληροφοριών προς τις δύο κατευθύνσεις. Ενδιάμεση, μέτοχοι, τράπεζες κλπ. Όλοι αυτοί παίζουν ένα ρόλο. Δεύτερο, και για να είμαι ειλικρινής, και είμαι ειλικρινής άνθρωπος, από την οικονομική άποψη αυτό και από την άποψη της ανταγωνιστικότητας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της πρότασης και αναφέρεται στην διαφάνεια μεταξύ θεσμικών επενδυτών και asset manager, αυτών που διαχειρίζονται δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία. Πάλι συχνά οι επενδυτές αυτοί είναι συνταξιωτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείε που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια, καμιά φορά και δημόσιου χρήματος. Είναι σαφές ότι απουσιάζουν συχνά αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες ευθύνες τους και δεν προσφέρουν επαρκή κίνητρα στους asset manager να στοχεύσουν και σε μακροπρόθεσμη απόδοση. Παράδειγμα, αν χρειάζεται να υποβάλεις ανατρίμηνο αναφορά για την απόδοσή του ως asset, απόδοσή σου ως asset manager, αυτό βεβαίως είναι πολύ βραχυπρόθεσμο και λαμβάνει υπόψη διάφορου δείκτε τη αγορά ανατρίμηνο ή εξάμηνο και επομένω στην ουσία σε αποθαρρύνουν να κοιτάξει και λίγο πιο μακριά. Αυτό που προτείνουμε εμεί λοιπόν είναι μια δέσμη μέτρων διαφάνεια. Όχι ούτε βαριέ διαδικασίε ούτε γραφειοκρατία. Διαφάνεια. Δείξτε ακριβώ τι κάνετε ω θεσμικό επενδυτή. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική σα. Ποιε είναι οι συμμαχίε σα και πώς συμβάλλεται στην μακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών σας στοιχείων. Δείξτε επίσης και ποια διασύνδεση υπάρχει μεταξύ του θεσμικού επενδυτού και του διαχειριστού των περιουσιακών στοιχείων, του asset manager, και πώς λειτουργούν αυτοί υπέρ του μακροπρόθεσμου συμφέροντος του επενδυτού. Και τέλος, ζητούμε από τους asset manager να αποκαλύπτουν στους επενδυτές ορισμένα πράγματα. Πώς διαχειρίζουν τα χρήματά τους, ποια είναι η απόδοση, ποιο είναι το κόστος. Διότι συχνά πολλές μελέτες δείχνουν ότι το κόστος ακόμα και αν είναι 0, κάτι μπορεί να είναι πολύ ψηλό. Διότι όταν έχετε ένα πολύ μακρό χρόνο απόδοσης, 30 χρόνια ας πούμε, για την ε, επένδυσή σε σύνταξη, μπορεί να είναι το ποσό τελικά πάρα πολύ μεγάλο. Σε ό,τι αφορά του ε, συμβούλου, όπω είπα προηγουμένως, proxy advisors, αυτοί βεβαίω παίζουν ρόλο στην συμπεριφορά, στην ψηφοφορία. Το τελευταίο, ε, η τελευταία τελεία τώρα. Αυτοί έχουν κώδικα διοντολογία. Καλώ. Εμά μας ικανοποιεί αυτό. Και είμαστε υπέρ βεβαίω του κώδικα διοντολογία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι χρειάζονται χρειάζεται να θεσπιστούν ορισμένε βασικέ αρχέ στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιδίω δύο πράγματα. Πρώτο, να είναι πολύ πιο ανοιχτή για το πώ φτάνουν στι συστάσει που κάνουν μετόχου να τηρήσουν μια στάση στην ψηφοφορία και δεύτερο πώ αντιμετωπίζουν τι συγκρούσει συμφερόντων, διότι εδώ πρόκειται για επιχειρήσει, οι οποίε χορηγούν συμβουλέ για την ψηφοφορία, αλλά χορηγούν συμβουλέ και για άλλα θέματα σε επιχειρήσει. Το άλλο θέμα, μέγα θέμα, είναι οι αμοιβέ. Αυτά λέχθηκαν και πριν από ορισμένους δικού σας. Εδώ συμφωνώ 200% με αυτά που λέει ο εισηγητής. Οι αμοιβέ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της επιχείρησης. Και βεβαίως αυτό είναι και το μακροπρόθεσμο ε, συμφέρον των μετόχων. Τρεις συστάσεις έχει κάνει στο παρελθόν η Κομισιόν για να βελτιωθούν τα πράγματα εδώ, αλλά βεβαίως τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά, όπως τα βλέπετε, τα διαβάζετε και στις εφημερίδες. Τι προτείνουμε τώρα, απλό πράγμα είναι, και μάλιστα είναι δύο απλά πράγματα. Πρώτο, εκ των προτέρων, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ψηφίζει πάνω σε μια πολιτική αμοιβών. Πώς θα πληρώνουμε δηλαδή το στελεχικό μας δυναμικό για τα επόμενα τρία χρόνια, με ποια κριτήρια απόδοσης, ποια θα είναι τα ανώτατα όρια των αμοιβών, όλα, όλα αυτά τα σχετικά δηλαδή. Αυτά όλα εκ των προτέρων και μετά, μετά από ένα χρόνο να υποβάλλεται έκθεση από την επιχείρηση για να δείξει τι έγινε. Έτσι λοιπόν, εκ των υστέρων, θα γίνεται, να, θα γίνεται ένα αφορά που θα λέει, κοιτάξτε, να, αυτό έγινε, αυτά πληρώνεται. Και νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα επεκτείνουμε και στην υπόλοιπη ε, αγορά. Αυτή είναι βασικά η, ιδέα. Μπορούμε να επιστρέψουμε αν θέλετε σε αυτό, αν θέλετε αργότερα. Τώρα οι συναλλαγέ με συγγενή μέρη. Και εγώ χρειάστηκε να κοιτάξω πρώτα τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει βασικά related party transactions ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν συναλλάσσονται μόνο στην ελεύθερη αγορά. Μπορούν να προβαίνουν και σε συναλλαγές μεταξύ της επιχειρήσεως και των διευθυντών της για παράδειγμα. Ή της οικογένειας που ε, διατηρεί στην κατοχή τη μεγάλο μέρος των μετοχών και θέλει για παράδειγμα να αγοράσει ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία τη εταιρεία. Τα λέω αυτά ως απλά παραδείγματα. Αυτά είναι, έχουν καλώς εφόσον γίνονται σε τιμές της αγοράς. Επειδή λοιπόν πρόκειται για συγγενές μέρος δεν είναι τόσο σαφέ αυτό ότι είναι τιμέ τη αγορά. Ω απλό μέτοχος ή ω μέτοχος μειοψηφία με ενδιαφέρει να γνωρίζω ότι οι συναλλαγές αυτές γίνονται σε τιμές της αγοράς, διότι τελείως υπονομεύεται η αξία της επενδύσεώς μου. Τώρα εδώ μπορεί να πει κανείς διάφορα πράγματα. Πρώτα εδώ υπάρχει έλλειψη πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Και υπάρχει πολλή υποστήριξη από πολλές μεριές για να δημιουργηθεί αυτή η διαφάνεια. Και το δεύτερο είναι τι γίνεται με σημαντικές τέτοιες συναλλαγές. Αυτό προτείναμε και εμείς. Άρα ψηφοφορία στην συνέλευση των μετόχων για τις πολύ μεγάλες συναλλαγές. Αυτό να γίνει είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων. Αυτό συζητείται ακόμα. Δεν θα σας κρύψω ότι στο Συμβούλιο το ζήτημα αυτό έχει προχωρήσει πολύ. Και όντως, όπως λένε στα αγγλικά, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πολλή δουλειά. Αλλά πάντως τη βασική αρχή νομίζω την δέχονται όλοι. Θα χρειαστεί λοιπόν περισσότερη διαφάνεια, περισσότερες ε, περισσότερη έλεγχη για τέτοιου είδους ε, μεγάλες συναλλαγές. Τέλος, ήδη στη νέα Κομισιόν ισχύει ένα περιβάλλον καλύτερης νομοθεσίας, better regulation. Δεν θα τα λέμε εκ των άνω λοιπόν. Πολλές από τις διατάξεις είναι πάνω σε βάση συμμόρφωσης ή εξήγησης comply or explain. Όταν μιλείτε για corporate governance υπάρχουν βεβαίω μεγάλες διαφορές εάν είσαστε στην Ιταλία, στην Αυστρία, στη Δανία. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη αυτές οι διαφορές των ε, χώρων μελών, εφόσον βέβαια εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο. Εγώ θα σταματήσω εδώ, αλλά δίπλα μου έχω τη συνάδελφό μου και αν θέλετε να της δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για αυτή την τόσο καλά δομημένη και πλήρη παρουσίαση. Μου λένε ότι θα είναι και διαθέσιμη στο διαδίκτυο η παρουσίασή σας, οπότε μπορούμε να την εξετάσουμε στη συνέχεια με πιο πολλή λεπτομέρεια. Έχετε να θέσετε κάποια ερωτήματα, να κάνετε κάποια σχόλια. Κυρία Ρέγκνερ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας έχετε τονίσει πάντα και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό ότι δεν πρόκειται μονάχα να αντιμετωπίσουμε μόνο το βραχυπρόθεσμο επίπεδο αλλά να δούμε και ποιο είναι το προσποριζόμενο όφελος για την εταιρεία, για την γενική κοινωνία, για τους καταναλωτές, για τους εργαζόμενους, να δούμε δηλαδή τη μακροχρόνια υγεία και στρατηγική μιας επιχείρησης. Έχω εδώ ένα πολύ βασικό ερώτημα. Λέτε ότι πρώτα απ' όλα να δούμε τη, τα πριμ και τους μισθούς των ε, στελεχών, γιατί προφανώς είναι ένα κίνητρο για αυτούς, αλλά αν εμείς δούμε μονάχα τα πράγματα από την οπτική γωνία των μετόχων, οι οποίοι φυσικά είναι και αυτοί εμπλεκόμενοι, νομίζω ότι αυτοί τους ενδιαφέρει ώστε να να είναι υψηλότερη η αξία των μετοχών τους. τότε με τον τρόπο και αυτό ενισχύεται αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη, να προσπαθούν μεγαλύτερο κέρδος στα, στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Μήπως είναι πάρα πολύ λοιπόν στενή η εστίασή σας σε αυτή την περίπτωση. Αν εμείς δίνουμε έμφαση στα δικαιώματα των ε, μετόχων, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα συμφέροντα των άλλων εμπλεκομένων. Αναφέρατε το explain or comply. Έχουμε όμως πολύ διαφορετικές δομές επιχειρήσεων στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εγώ υπήρξα εισηγήτρια για το Women on Board, για τη συμμετοχή των γυναικών στα εταιρικά συμβούλια. Εδώ ε, λειτουργήσε αυτή η, η αντιμετώπιση του comply or explain. Σε άλλες περιπτώσεις όμως όχι. Πώς λοιπόν μπορούμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ε, μετόχων, αλλά παράλληλα και τα δικαιώματα να ενισχύσουμε των εργαζομένων και των καταναλωτών όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε μια επιχείρηση και πώς ακριβώς θα το επιτύχετε αυτό με τη διαδικασία comply or explain. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα για τις λεγόμενες related party transactions, για τις συναλλαγές ε, σχετιζόμενων συμβαλωμένων. Εδώ υπάρχει το θέμα του να υπάρχουν ανεξάρτητες κρίσεις και τα λοιπά. Μήπως όμως αυτό θα οδηγήσει και σε μια αύξηση της γραφειοκρατίας, όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε με την καλύτερη ρύθμιση δεν θα εξανεμιστούν. Μήπως ε, μια επιχείρηση δεν θα ήταν καλύτερο να μπορεί να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις διαδικασίες χωρίς περισσότερη γραφειοκρατία και όταν αυτά πρέπει να έρθουν στην ε, Γενική Συνέλευση, τι γίνεται με τα απόρριτα τα οποία θα πρέπει να αποκαλυφθούν σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται η σύγκληση της συνέλευσης των μετόχων και τι πρόσθετο κόστος μπορεί να ε, σημαίνει αυτό ότι θα υπομειστεί μια επιχείρηση. Και τέλος, σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα συναπόφασης μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Αν αποφασίζει η συνέλευση λοιπόν των μετόχων και παρακάμπτει κατά κάποιο τρόπο αυτό την συναπόφαση των εργαζομένων, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Ζεμπετών. Αυτό το σχέδιο τροποποίησης είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι και κάπως συμπαθητικό, διότι τελικά δίνει μια ηθική χρειά στον καπιταλισμό, να δώσει ηθικό στον καπιταλισμό και θέλει να καταστήσει το καθεστώς αυτό με επενδυτικό καπιταλισμό. Θα είναι δύσκολο το έργο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη και αυτή στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Η παγκοσμιοποίηση δεν εξηγεί τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεθάρρυνε μια πολιτική υπερβολικά φιλελεύθερη, ευνόησε κατά πολύ τη δυνατότητα μετακίνησης διακίνησης κεφαλαίων, ευνόησε συνεπώς αυτό το χρηματιστικό και ε, καπιταλισμό που έδωσε τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε. Τα στοιχεία που παρετέθησαν 72% των μετοχών πολλούνται κάθε χρόνο. Είναι τρομακτικός αυτός ο αριθμός. Αντί να συναγάγουμε συμπεράσματα από αυτό, εξακολουθούμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αποδυναμώνουμε τις χώρες, μειώνουμε την εθνική προστασία, ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι πρέπει να καταργήσουμε την γραφειοκρατία. Αυτό πώ ερμηνεύεται εθνική προστασία. Ε, εδώ σε αυτό το θεσμικό όργανο υπάρχουν γραφειοκρατία, σημαίνει προστατευτισμό εθνικό που θα πρέπει να καταστρέφεται συνεχώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τι χώρε εναντί τη αγορά, τι χώρε που αποδυνάμωσε αφήνει ελεύθερο το χώρο στις πολυεθνικές, στα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν λίγο πολύ. Οι πολίτες ε, μένουν σαν τους παρτιάτες που πολεμούν χωρίς καμία θωράκιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σαν πυρομανής πυροσβέστης που θέλει να σβήνει τελικά τις πυρκαγιές που ήδη ανάβει. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόιερ μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά που υπόθηκαν. Λοιπόν, να τα συναθρήσουμε όλα αυτά. Η κυρία Ρέκνερ αναφέρθηκε στην ενίσχυση των μετόχων. Είναι σοφό αυτό. Μήπως πετυχαίνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το ερώτημά σας. Από τις συνομιλίες μας και τις συζητήσεις ε, καταλήξαμε στο να συζητάμε τους μεγάλους μετόχους. Και υπάρχει και ένα συνέστημα ευθύνης ε, για εκείνους που διαχειρίζονται μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιδοτικά ταμεία που διαχειρίζονται χρήματα για μας και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν όπως σήμερα και στο μέλλον. Δεύτερον, όλο και περισσότερο υπάρχουν θεσμικοί επενδυτές, μάλλον επενδυτές που εξετάζουν θέματα διακυβέρνησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Αυτοί οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία και αλλού καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από το κέρδος, αλλά και η οπτική γωνία η μελλοντική του περιβάλλοντος, κοινωνικές πτυχές κλπ. όταν χειρίζονται, διαχειρίζονται μια επιχείρηση. Αυτή είναι οι φορείς που θα πρέπει να επεξεργαστούμε και να σας πω ότι σε κάποια κράτη-μέλη, σε αρκετά κράτη-μέλη, αυτό το σχήμα όπου αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες οι μέτοχοι και έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και έχουν περισσότερες δυνατότητες, λαμβάνει ήδη χώρα σε κάποια κράτη-μέλη. Στη χώρα μου, στην Ολλανδία, είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Έχω την πεποίθηση λοιπόν ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και όσοι έχουν τα πράγματα τώρα ε, δεν υπάρχει και εναλλακτική όσον αφορά και την ε, αυτό συμμόρφωση εξήγηση, comply or explain. Αυτό δεν, δεν λειτουργεί πάντα, πράγματι. Γι' αυτό είναι ένα μοντέλο συμμορφώσου ή εξήγησε, comply or explain. Ε, είναι ένα πλαίσιο υπείου δικαίου. Υιοθετήσαμε τον Απρίλιο ε, μια σύσταση που αφορά την εξήγηση. Λένε οι επιχειρήσεις δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε αλλά μας λείπει η εξήγηση. Και αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σύσταση είναι καλός, ε, γίνεται αυτό. Εξηγήστε όμως ποια εναλλακτική θα ακολουθήσετε, για πόσο χρόνο ε, και πώς θα πετύχετε τελικά τον βασικό στόχο της ε, νομοθεσίας. Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε την πλευρά της ε, εξήγησης και θα μας ενημερώσουν σε κάποια φάση τα κράτη-μέλη πώς εφαρμόζουν το Comply Explain αυτό το μοντέλο, αλλά αφορά ήπια νομοθεσία για την ώρα. Όσον αφορά τις συναλλαγές ε, των ε, συμβαλωμένων μερών, των σχετιζομένων μερών, δεν ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, διότι είναι τεχνικής φύσεως η πρόταση. Νομίζω ότι όπως προανέφερα όμως, κατανοήσαμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην δυσχεράνουμε την κατάσταση, να μην βλάψουμε εμπορικά βιομηχανικά ε, συμφέροντα ή να μην αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Επεξεργαζόμαστε και θα ενημερώσουμε τον εισηγητή με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Ο στόχος όμως είναι κοινό για όλους. Δηλαδή η μειοψηφία των μετόχων δεν θα πρέπει να υποφέρει Δηλαδή ότι αυτοί που έχουν εσωτερική γνώση μπορούν να συναλλάσσονται με τις επιχειρήσεις και να ε, επηρεάζουν το καθεστώς ιδιοκτησία εκείνων που είναι εκτός. Ε, σημαντικότατος ο στόχος πώς μπορεί να επικρατεί σωστή διαφάνεια και να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ διαφάνειας ε, και να μην αυξήσουμε το άχθος. Αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα, θα το εξετάσουμε. Τέλος δεν είμαι σίγουρος εάν κατανόησα την ερώτηση, την τελευταία, αν την ερμηνεύω σωστά, να το πω με δικά μου λόγια. Εδώ δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον καπιταλισμό ή την κοινωνία. Ε, προσπαθούμε ε, να καλύψουμε κάποιες εντοπιστήσεις αδυναμίες και προσπαθούμε να έχουμε πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων δεν αφορά τόσο καθαρά αριθμητικά στοιχεία. Αφορά περισσότερο το πνεύμα, την προσέγγιση. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές πτυχές, τα συμφέροντα άλλων εμπλεκομένων μακροπρόθεσμα ζητήματα. Αν είναι 70, 40, 50% αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Τελικά, Πρόεδρε, κλείνοντας, Πρέπει να πω ότι ξέρω ότι και στο Κοινοβούλιο πολλοί ενδιαφέρονται πολύ για τις αμοιβέ, για τις πληρωμές και διαβάζουμε διάφορα άρθρα στον τύπο πόσο ε, υψηλή είναι η μισθή και οι έκτακτες αμοιβέ, τα μπόνουσες. Το σημαντικότερο όμως είναι η μεγάλη, να έχουμε σωστή σχέση μεταξύ μεγάλων θεσμικών επενδυτών και ε, των αμοιβών των στελεχών. Εδώ βρίσκονται ε, τα πολλά χρήματα, ε, εκεί προστατεύονται ή μάλλον αυτά είναι που αφορούν τα βασικά συμφέροντα της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πρόεδρος για τις απαντήσεις. Μέσω της σημαντικής συζητήσεως αυτής μείναμε λίγο πίσω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Αν συμφωνούν λοιπόν τα μέλη, ας ακολουθήσουμε την παράδοση της Επιτροπής να ψηφίζουμε συγκεκριμένη ώρα αν επιτρέπει λοιπόν η Επιτροπή για την ώρα θα αφήσουμε το σημείο 12 η παρουσία σε πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τροποποίησης ε, της διαδικασιών ε, recast και ας πάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες, στα σημεία των ψηφοφοριών. Θα ξεκινήσουμε από το 13 Και το λόγο έχει η συγγήτρια η κυρία Χαουτταλά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι επίμαχη η έκθεση, δεν υπευλήθησαν τροπολογίες, όπως, οπότε συστήνω στην Επιτροπή να στηρίξει αυτή τη σύμβαση. Ε, ευχαριστώ. Είμαστε στο σημείο 13 και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τώρα τις κάρτες ψηφοφοριών, όπως μου λέγουν. Παρακαλώ πάρτε τις κάρτες σας και παρακαλώ να βάλτε τις κάρτες σας στα μηχανήματα. So, uh, the Λοιπόν, η συγγήτρια είναι να υθετήσουμε την ε, πρόταση και ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Εψήφισαν 20, 18 ψήφοι υπέρ, 2, 2 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Πάμε στο σημείο 14. Η συγητή είναι υποφαινόμενο. Να πω τη σύμβαση της Χάγης του 2005 για τις συμφωνίες για επιλογή δικαστηρίων αφορά ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και σχετικά θέματα αφορά αποκλειστική επιλογή ε, δικαστηρίων σε θέματα εμπορικά και ιδιωτικά. Σκοπός της συμβάσεως είναι παρόμοιος με το άρθρο 25 του κανονισμού Βρυξελών 1 ε, του αναδιατυπωθέντος βασική χρήση της συμβάσεως εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για διεθνή απο... για συμφωνίες διεθνής αποκλειστικής επιλογής δικαστηρίων, οπότε τονώνει και τη συνεργασία συμμετοχών των κρατών μελών. Έχει επικυρώσει τη συμφωνία μόνο το Μεξικό, αλλά συνεχίζονται οι σχετικές διαργασίες στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω το Κοινοβούλιο να δώσει σύμφωνη γνώμη στην απόφαση του Συμβουλίου που κυρώνει την σύμβαση. Υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να σχολιάσει πριν προβούμε στην ψηφοφορία. Ουδέν σχόλιον. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Η εγκρίνεται, εψήφισαν 20, 18 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Πάμε τώρα στο σημείο 15 έως 28. Ο κύριος Ντούντα μπορεί να σχολιάσει όλα τα σημεία μαζί. Αν επιθυμεί να προβεί σε κάποια σχόλια. Ο κύριος Ντούντα είναι εδώ. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση μπορούμε να ψηφίσουμε όλα αυτά τα σημεία μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίσαντες 21. Υπέρ 19. Δύο αποχές μηδέν ψήφοι κατά εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. Ε, Πάμε στο σημείο 41 έγκριση σχεδίου γνωμοδοτήσεως υπομορφή επιστολής όσον αφορά αναφορά 1784 κάθετος 213-2013 Τζιλμπέρτι για κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Το σχέδιο επιστολής έχει διανεμηθεί. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε. Αρκεί να ψηφίσουμε διανατάσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές Δύο εποχές. Καλώς εγκρίνεται. Ε, by special request we... Με ειδική αίτηση ζητούμε, μας ζητήθηκε να ψηφίσουμε την, ε, τον αριθμό 30. 30 με 32 και δίνω το λόγο στην κυρία Γκέρνγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να παρουσιάσω την έκθεση σε σχέση με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οποία τροποποιεί τον κανονισμό 861 κάθετος 2007 της 11ης Ιουλίου 2007. Ο κανονισμός αυτός θεσμίζει τη διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών. και επίσης του κανονισμού 1896 κάθετος 2006 12 Δεκεμβρίου του 2006 που θεσπίζει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Πληρωμών. Έχω ήδη υποβάλει ένα έγγραφο εργασίας και τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω το σχέδιο της έκθεσής μου. Εν γέννη, πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ καλή και γι' αυτό πρότεινα μονάχα ορισμένε τροπολογίες οι οποίες κάνουν πιο εξειδικευμένη αυτή την πρόταση. Για το γενικό πλαίσιο τώρα. Έχουμε μια οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε βελτίωση στην ε, αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του δικαίου θα υποστηρίξει την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεών μας και την ανάκαμψη. Οι τροπολογίες σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών οδηγούν σε αυτό το στόχο. θέλω να σας δώσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την χρήση αυτού του εργαλείου το οποίο εφαρμόστηκε το 2007. Λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε με μη ικανοποιητικό τρόπο. Γιατί το κατόφλι ήταν πολύ χαμηλό, ήταν μονάχα 2.000 ευρώ. Και η διαδικασία αντιμετωπίστηκε από τους καταναλωτές ως μια επαχθής διαδικασία, μια χρονοβόρα διαδικασία και δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη διαδικασία αυτή η οποία θα μπορούσε να ελαφρώσει το έργο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Συστήματος και δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής η διατάξεις της. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο 12% αυτών οι οποίοι έτυχαν ε, σφιγμομέτρησης γνωρίζαν ότι υπήρχε αυτό το εργαλείο και ξέρανε ποιες ήταν οι δυνατότητές του. Και μόνο 1% <clears throat> αυτών των ιδίων χρησιμοποίησε πράγματι αυτή τη διαδικασία διευθέτησης μικροδιαφορών. Κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο σε διαμεθοριακές υποθέσεις θα ήταν το να μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία γραπτός, χωρίς εμφάνιση στο δικαστήριο και την προσφυγή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Θα ήθελαν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επιγραμμική πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία και να χρησιμοποιούν και τη μητρική τους γλώσσα. Και αυτά ήταν τα πιο σημαντικά στοιχεία στην έρευνα της Κομισιόν. Ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε. Καταρχήν να διευρύνουμε τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού σε διαφορές που φτάνουν μέχρι και 10.000 ευρώ ε, και όχι μόνο 2.000 σε διαμεθοριακές περιπτώσεις. Όχι μονάχα για μεμονωμένους κατανάλωτες, αλλά και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προτείνουμε λοιπόν να διευρύνουμε και την έννοια των διαμεθοριακών υποθέσεων και να χρησιμοποιήσουμε και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για την υποβολή εγγράφων επίσης. Τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν βιδεοδιασκέψεις και άλλες μορφές επικοινωνίας ώστε να διεκπαιρεωθεί ταχύτερα η διαδικασία στα δικαστήρια. Δεν είναι όμως ε, ε, εξοπλισμένα όλα τα δικαστήρια με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις πληροφορικές λύσεις. Πιστεύω ότι επομένως αυτό θα πρέπει να γίνει να εξασφαλιστεί δύο χρόνια μετά τη θέση εφαρμογή αυτού του νέου νομοθετήματος. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι υπάρχει και ένα λογικό επίπεδο τελών δικαστηριακών. Σε ορισμένε περιπτώσεις τα δικαστικά τέλη ήταν τόσο υψηλά που δεν είχε και νόημα να κάνει κανείς μια αγωγή διότι το κόστος της δικαστικής διαδικασίας θα υπερεύαινε το προσποριζόμενο κέρδος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, προτείνουμε τα δικαστικά τέλη να πληρώνονται εξ αποστάσεως. Γιατί σε πολλές χώρες, σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να πάει κανείς αυτοπροσώπος και επιτοπίως να πληρώσει τα δικαστικά τέλη με ένα με ειδικό ένσημο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πληρώνονται με πιστοτική κάρτα, με τραπεζική ε, επιταγή και ένας άλλος τρόπος για να μειωθεί το κόστος της διαδικασίας θα ήταν να περιοριστεί η ανάγκη μετάφρασης ε, και να γίνεται μετάφραση μονάχα για τα έγγραφα που αναφέρονται στο παράδειγμα Δέλτα. Δεν χρειάζεται να μεταφράζονται όλα τα έγγραφα για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει η δικαστική απόφαση και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους. Βάσει της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαφορές ύψους 2 έως 10.000 ευρώ θα αντιπροσώπευαν το 30% όλων των διαφορών. Περίπου το 1 πέμπτο των ε, διαφορών που έρχονται στα δικαστήρια θα ξεπερνούσαν το ύψος των 2.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμα μία τροποποίηση. Μία τροπολογία που θέλω εγώ να προτείνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα κατόφλι σε σχέση με το αίτημα η δικαστική διαδικασία να γίνει στην πράξη. Να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Η διαδικασία ε, μικροδιαφορών γίνεται κανονικά με γραπτή διαδικασία. Αν δεν μπορεί όμως το δικαστήριο να εκδώσει μια απόφαση επί τη βάση των στοιχείων των γραπτών που έχουν δώσει τα δύο αντίδικα μέρη ή αν ένας αντίδικος ζητήσει να υπάρξει προφορική διαδικασία, τότε θα πρέπει να γίνει μια επίσημη δίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρχει εδώ ένα κατόφλι 2.000 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις όταν η μία από τις δύο πλευρές ζητά να υπάρξει προφορική διαδικασία. Εγώ προτείνω να φτάσει στα 5.000 ευρώ αυτό το όριο, το κατόφλι, με την προϋπόθεση επίσης ότι θα υπάρξει συμφωνία και των δύο πλευρών για να ε, φτάσουν στα δικαστήρια εφόσον έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας επί τη βάση της γραπτής διαδικασίας. 5.000 ευρώ θα χρειάζεται λοιπόν για να γίνει προφορική διαδικασία. Εγώ Υποστηρίζω ιδιαίτερα αυτόν τον νέο κανονισμό για την άποψή μου θα είναι πολύ αποτελεσματικός αλλά δεν θα μπορεί να ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πρόκειται για τροπολογίες ενός κανονισμού που ήδη ισχύει αλλά δεν καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη αυτού του κανονισμού και αυτά ήθελα να σας πω. Μόναχα ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με το ανώτατο όριο των δικαστικών τελών. Πιστεύω ότι το κόστος της διαδικασίας δεν θα ξεπερνάει το 10% της επίδικης αξίας ώστε να αξίζει τον κόπο για τους ε, διάδικους να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Επίσης έχω συμπεριλάβει και μία σύσταση προς τα κράτη-μέλη σε σχέση με τη δυνατότητα να μην υπάρχουν δικαστικά τέλη για άτομα τα οποία, για διάδικους οι οποίοι έχουν μονάχα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Αυτά λοιπόν. Η έκθεσή μου είναι μονάχα στα αγγλικά διαθέσιμη προς το παρόν. Καλύπτει όλες αυτές τις προτάσεις που σας προανέφερα και προσβλέπω στις προτάσεις και τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω κάτι ενημερωτικά. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την έκθεση είναι 27 Νοεμβρίου. Σημειώστε το σας παρακαλώ. Θέλει κανείς να πει κάτι. Ε, Mr. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίασή της, για την έκθεσή της Συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις της. Χαίρομαι που τα βασικά στοιχεία της ε, προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μετεβλήθησαν. Τι ο τρόπος η πρόσβαση δικαιοσύνη θα βελτιωθεί, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρές διαφορές για την ώρα ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού και τώρα μεγαλύτερος αριθμός ε, πιστωτών θα έχει πρόσβαση σε αυτή την ε, επίλυση των διαφορών και έτσι θα διευκολυνθεί και η διακίνηση κεφαλαίου και θα ενθαρρυνθεί και το διασυνοριακό εμπόριο και θα λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά. Ε, δύο στοιχεία θα ήθελα να προσέξουμε αυξάνοντας το κατόφλιο πρώτα απ' όλα από 2.000 στα 5.000 ευρώ, αυτό θα μειώσει το κόστος των διαδικασιών, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι τα δικαιώματα των διαδίκων διαφυλάσσονται. Δεύτερον, ο περιορισμός του τρόπου πληρωμών που προβλέπεται από τα δικαστήρια. Μόνο μια επιλογή ουσιαστικά προβλέπεται. Είτε τραπεζικό έμβασμα ή πληρωμή με πιστοτική κάρτα. Νομίζω ότι έτσι αυξάνονται οι δυσκολίες για τους πολίτες. Καλύτερο είναι να υπάρχουν περισσότερες επιλογές στην πληρωμή. Αν κάποιος δεν έχει πιστοτική κάρτα, φέρει πίν, και είναι η μόνη επιλογή που προβλέπει το δικαστήριο, που επιτρέπει το δικαστήριο, πώς θα πληρώσει. Βέβαια, ίσως να χρειαστεί κάποιος χρόνος να εισαχθούν και άλλες ε, μορφές πληρωμών. Όμως, θα μπορούσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία γι' αυτό. Όπως ίσως θα μπορούσε να επεκταθεί και μια χρονική περίοδος που προβλέπει την, την χρήση βίντεο διασκέψεων. Ο κύριος Φως έχει το λόγο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ εντατικά ακόμη με το θέμα. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι το στοιχείο αυτό είναι κατ' επιλογή, είναι προαιρετικό. Μπορώ να ακολουθήσω και τη συνήθη νομική οδό. Ή είναι υποχρέωση. Εφόσον υπάρχει απέτηση μέχρι 10.000 ευρώ. Και η άλλη ερώτηση τώρα, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει κατ' επιλογή, είναι προαιρετικό άρα, υπάρχει όμως και ο παραδοσιακός τρόπος έως το ύψος των 10.000 ευρώ, Ίσως αυτός λοιπόν ο παραδοσιακός τρόπος είναι και πιο ασφαλής. Γιατί για πολλούς τα 10.000 ευρώ δεν είναι βεβαίω και καμία περιορισμένη απέτηση, καμία χαμηλή απέτηση, είναι υψηλή. Το ζήτημα είναι λοιπόν, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ηλεκτρονική διαδικασία, μήπως προτιμούν να εκπροσωπηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Το άλλο είναι τα γλωσσικά κολλήματα. Αν πάω εγώ τώρα στη Φιλανδία για παράδειγμα και θέλω να προβάλλω μια απέτηση, είμαι υποχρεωμένος να ε, το κάνω αυτό στα φιλανδικά, διότι βεβαίως οι κανονισμοί των δικαστηριών λένε πάντα ότι η επίσημη γλώσσα είναι η γλώσσα του κράτους όπου έχει την έδρα το δικαστήριο. Βλέπω κάποια προβλήματα εκεί για το συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Τώρα για την τηλεμετάδοση, τη βιντεομετάδοση. άψη διαδικαστική, δικονομική διαδικαστική. Γίνεται αυτό στις διάφορες χώρες μέλη. Μήπως πρέπει να γίνουν προσαρμογές στους κανονισμούς των δικαστηρίων και τι γίνεται με τις τεχνικές υποδομές και τι γίνεται εάν διακοπεί η μετάδοση. Τι γίνεται με, τα, με τις προθεσμίες ή με τα κολλήματα, με τις απουσίες δηλαδή δικαιολογημένες απουσίες κάποιων ε, διαδίκων. Δεν πρέπει εκεί να σκεφτείτε λίγο τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και αυτά που είπε ο κύριος Άρντεφ προηγουμένως. Τα τέλη των ε, εμβασμάτων μέσω πιστοτικών καρτών. Πάλι εδώ νομίζω ότι στις διάφορες χώρες μέλη, στις διάφορες χώρες τα τέλη είναι διαφορετικά για τις διάφορες διαδικασίες. Και εκεί λοιπόν η ερώτησή μου είναι μήπως αυτό έχει μεταγενεστέρως κάποιες επιπτώσεις. Ξανοίγομαι λίγο περισσότερο τώρα σε διαδικαστικά ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι συνεπάγονται αυτές οι ρυθμίσεις και γι' αυτό επιστρέφω στο κέριο ερώτημα, είναι υποχρεωτική αυτή η διαδικασία ή είναι κατ' επιλογή, όπου μπορεί κανείς να αποφασίσει είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο κ. Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να εισαρώ την εισηγήτρια για το έργο της. Χρειάστηκε πολλής χρόνος, μεγάλες προσπάθειες, αποδοτική προσόγγιση. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άκρο ευπρόσδεκτη για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Διότι θα διευκολύνει τις ε, διασυνοριακές αξιώσεις. Και ένα από τα αποτελέσματα θα ήταν η επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και η απλούστευση των διαδικασιών για τα δικαστήρια. Εάν είναι γραπτή διαδικασία θα είναι υποφελής για τα δικαστήρια. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι που σχετίζεται με τη δυνατότητα αύξησης του ανωτάτου ορίου όταν αναφερόμαστε στις μικρομεσές επιχειρήσεις. Διότι τα ποσά με τα οποία ασχολούνται είναι υψηλότερα από εκείνα που χρησιμοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα. Μπορούν να φτάσουμε και 15.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Βος, κατά πόσο είναι υποχρεωτική ή όχι η διαδικασία ή αν είναι δυνητική. Νομίζω ότι το κείμενο προσφέρει επαρκή εχέγγυα ούτω ώστε τα δικαιώματα εκείνων που χρησιμοποιούν τη διαδικασία να είναι προστατευμένα. Διότι αναφέρεται ρητά ότι η αξίωση είναι πάνω από 5.000 ευρώ τότε είναι υποχρεωτικές οι προφορικές συζητήσεις και τα μέρη έχουν τα, το δικαίωμα να ζητήσουν με τέτοια προφορική συζήτηση και έτσι καλύπτονται τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα, αφορά όλους. Σχετίζεται με τη διαβίβαση των πληροφοριών στο δημόσιο χώρο, ούτως ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορούν να ακολουθούν την απλουστευμένη διαδικασία. Ίσως θα πρέπει η διαβίβαση των πληροφοριών να εξεταστεί, ούτω ώστε οι πραγματικοί δικαιούχοι να γνωρίζουν ότι υφίσταται αυτή η απλουστευμένη ε, διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρίνιο Εμπίντου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν λάβω το λόγο, πριν αρχίσω μάλλον να λαμβάνω το λόγο θέλω να αναφερθώ στις αμφιβολίες του κυρίου Άξελ Βος. Συμφωνώ και εγώ ότι πράγματι υπάρχουν αμφιβολίες και πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση. Υπάρχει ένα άλλο σημείο για το οποίο θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου, γιατί το θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η αξιοπρέπεια μιας δικαστικής διαδικασίας δεν πρέπει να εξαρτάται μονάχα από την οικονομική αξία η οποία διακυβεύεται. Και οι μικρές διεκδικήσεις, οι διεκδικήσεις χαμηλού ποσού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια αξιοπρέπεια όσο και οι μεγαλύτερες διεκδικήσεις. Δηλαδή η ακραία δικαστική απλοποίηση μπορεί να δώσει στις διεκδικήσεις αυτές ένα ίσον δικαστικό καθεστώς να δημιουργηθεί ένας ευτελισμός κατά κάποιο τρόπο της διαδικασίας και των εμπλεκομένων. Εγώ θεωρώ, τη χάρη, ότι δεν έχει νόημα να μην υπάρχει παρουσία δικηγόρου σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο δικηγόρος δεν είναι ένας οικονομικός παράγων ο οποίος θα αυξήσει την, το κόστος της διαδικασίας. Έχει ένα σημαντικό ρόλο ο δικηγόρος στο να εξασφαλίσει την ισότητα όπλων των διάδικων πλευρών. Οι πλευρές αυτές οι οποίες έχουν εκπροσώπηση μέσω δικηγόρου, συγγνώμη, έχουν μεγαλύτερη ισότητα έναντι του δικαστή. Στην περίπτωση που όμως μόνο μία από τις δύο πλευρές εκπροσωπείται από δικηγόρο ή δεν υπάρχει καμία παρουσία δικηγόρου, είναι πολύ μικρότερη η ισότητα και πολλές φορές δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των συμφερόντων κάθε πλευράς. Ακόμα και για μια υπόθεση χαμηλού οικονομικού ύψους θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση με δικηγόρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα ώστε όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα <clears throat> από την οικονομική τους ευρωστία και ιδίως όταν δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα που να τους επιτρέψει να προσλάβουν ένα, συνήγορο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία με μια ε, παροχή από την πλευρά του του κράτους αυτής της προστασίας. Ο κύριος Βίλαντ, θέλετε να πείτε κάτι. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική ψηφία, μια σημαντική ψηφίδα για το θέμα του δικαίου. Η καθυστέρηση δικαιοσύνης δεν είναι δικαιοσύνης, πρέπει να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα τώρα το αν πρέπει να υπάρχει παρουσία δικηγόρου ή όχι. Υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα κράτη-μέλη για το πότε μπορεί κανείς να έχει την αξίωση της παρουσίας ενός δικηγόρου και όταν δεν μπορεί κανείς να έχει την οικονομική αυτή δυνατότητα υπάρχουν ρυθμίσεις για την ε, πώς την αυτεπάγγελτη παρουσία δικηγόρου. Αλλά δημιουργούνται πολύ εύκολα προβλήματα με όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε την ε, ταχύτητα, ταχύτητα της διαδικασίας. Μπορεί να υπάρχει περίπτωση <clears throat> όμως όπου ε, κάποιος έχει πάρει παράδοση του αγαθού, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση αυτή πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μικρό διαφορά όταν ο, ο αγοραστής παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το οποίο του έχει παραδοθεί αλλά ο πιστωτής του έχει κάθε απόδειξη ότι έχει κάνει τα απαραίτητα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε διαδικασίες οι οποίες είναι ε, γρήγορες και θα μπορούν να λειτουργούν και σε διαμεθοριακό επίπεδο με αποτελεσματικό τρόπο. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να εξασφαλίσει την, ε, ε τίτλο, τον τίτλο αυτό, να εξασφαλίσει την παράδοση του τίτλου, ο οποίος δικαιολογεί την ανάγκη να υπάρξει μια πληρωμή. Χειρότερη περίπτωση είναι ο πελάτης ο οποίος ενώ πρέπει να πληρώσει δεν θέλει να πληρώσει ή δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτός ο κακόπιστος ε, τελικά ο φιλέτης είναι αυτός δηλαδή ο οποίος μπορεί να πληρώσει αλλά δεν θέλει να πληρώσει θα ψάχνει πάντοτε να βρει διαδικασίες για να ξεφύγει. Αυτό όμως εμείς πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί εκεί εντοπίζονται δυσκολίες που είπε ο κύριος Βόσ, αλλά και άλλοι. Πρώτα λοιπόν, πώς θα βοηθήσουμε τους καλοπροαίρετου συναλλασσόμενους να προχωρήσουν στη βάση μιας ε, διαδικασίας διασυνοριακής, η οποία θα επιτρέπει την ταχύτατη εξέλιξή της. Για όλα τα υπόλοιπα, είτε μπλέκεται δικηγόρο είτε όχι, μπαίνουν τα ζητήματα πώ θα βοηθήσω πρώτα τον οφειλέτη, πώ θα βοηθήσω τον ε, πιστωτή και ποιο θα δώσει τη λύση. Γιατί αλλιώ δημιουργούμε διαδικασίε με υψηλό κόστο. Και εκεί νομίζω το ξεφεύγουμε από τα όρια. Πρέπει κυρίως να εξετάσουμε τον καλής προθέσεως πιστωτή και τον καλής προθέσεως οφειλέτη. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας για την θέσπιση διαδικασίας και να βρούμε ξεκάθαρες απαντήσεις που να είναι μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπρούνι της ε, Ιταλικής Προεδρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα για μία ακόμη φορά σε όλους σας. Όπως είπε η συγγήτρια, θα ήθελα και εγώ να περιγράψω την κατάσταση από την πλευρά μας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του κειμένου. Όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο ακόμα το επεξεργάζεται. Πρόθεσή μας είναι να καταλήξουμε σε συμβιβαστικό κείμενο που θα υποβάλουμε στην Κορεπέρ την επόμενη εβδομάδα, ελπίζοντας ότι μετά μπορούμε να υποβάλουμε ε, το κείμενο στο Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου για γενική συζήτηση. Τον κανονισμό τον θεωρήσαμε πάντα σημαντικότατο και ήταν από τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Ο ίδιος ο κ. Υπουργό, ο κ. Ολάντο, όταν παρουσίασε το πρόγραμμα του στην Νομική Επιτροπή, ανέφερε ότι πρόκειται περί ενός μέσου που ακολουθεί την κατεύθυνση διευκόλυνσης της δικαιοδοσίας προς όφελος όλων των ε, εκείνων που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει και έμεση συνέπεια του κανονισμού. Δεν είναι καλό μέσο μόνο διότι εγγυάται μια ταχύτητα κυρίως όσον αφορά τις, ε, τους μικρούς φορείς και τις μικρές διαφορές αλλά έχει και έμεση συνέπεια να μειώσει το άχθος εργασίας των δικαστηρίων ε, που έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας ε, πολλά δικαστήρια σε πολλές χώρες λόγω των υποθέσεων. Τον κανονισμό τον συζήτησε και με κάποια ένταση το Συμβούλιο και εμπεριέχει στοιχεία σημαντικότατα. Θα είμαι λακωνικός, θέλω να αναφερθώ σε κάποιες προτάσεις που ακούστηκαν από τους ε, αξιότιμους βουλευτές το θέμα της χρήσης της τεχνολογίας. Είναι σημαντικότατο θέμα. Εμείς στο Συμβούλιο το θεωρούμε αυτό ότι είναι θετικό στο βαθμό στον οποίο βοηθά ε, πιο τακτική και ταχύτερη επίλυση των διαφορών. Δεν είναι ένα μέσο για να απομακρυνθεί ο τελικός χρήστης από τον δικαστή. Δεν υπάρχει πρόθεση να αφαιρέσουμε τη δυνατότητα από κάποιον διάδικο να έρθει επαφή με το δικαστή. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι και το εξής. Να τονίσουμε το πρόβλημα που ανέφερε ο κύριος Πίντου. Δηλαδή να υπάρχει να δώσουμε ε, νομική αξιοπρέπεια σε όλες τις αποφάσεις. Ακόμα και εκείνες που είναι αφορούν μικρότερα ποσά, μικρότερες διαφορές διευκολύνει ο κανονισμός και αυτή την πτυχή. Σαν Προεδρία ενδιαφερόμεθα πολύ να αφήσουμε ανοιχτή τη συζήτηση της διάβολης επικοινωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με χαρά άκουσα την παρουσίαση της συγγήτριας. Όσον αφορά το χρονισμό και τις περαιτέρω εξελίξεις, με τα χαρά να σας ενημερώσω ότι επεξεργαζόμαστε εντατικά το θέμα ούτως ώστε να πετύχουμε τη συνένεση των κρατών μελών εν ώψη του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014. Η θέση του Συμβουλίου είναι κοντά σε κάποια λύση, σε κάποια κατάληξη. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν σας δίνω λεπτομέρειες, διότι δεν έχουμε ακόμα ένα κείμενο και εφόσον δεν έχουμε κείμενο το θεωρώ πρόημο θα ήθελα να εκφράσω κάποια αισιοδοξία όσον αφορά το συγκεκριμένο όμως ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, Γιάτσεκ Γκάφσκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την παράκληση να είστε κάπως σύντομος, διότι έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με το πρόγραμμά μας, αρκετά πίσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία εισηγήτρια για το κείμενο αυτό, το σχέδιο κειμένου, ευπρόσδεκτο, ευπρόσδεκτες και όλες οι προτάσεις που εμπεριέχονται στο σχέδιο κειμένου. Αξίζει πιστεύω να θυμηθούμε ότι είναι δυνητική αυτή η διαδικασία, δεν αποκλείει και διάφορες εθνικές προβλέψεις. Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιταχύνει τις διασυνοριακές τέτοιες ε, επιλύσεις διαφορών και αφορά τις διασυνοριακές υποθέσεις και θα εξακολουθεί να έχει αυτή τη μορφή. Στόχος είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω απλούστευσης και μειώσεως του κόστους. Αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε ήδη για πέντε χρόνια και δεν ακούσαμε ποτέ καμία διαμαρτυρία. Δεν ισχυρίζεται και κανείς ότι δεν παρέχει τα αναγκαία χέγγια στα μέρη. Στην πρότασή μας βλέπετε αυξάνουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις εγγύσεις για τα διάδικα μέρη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ σύγχρονη διαδικασία και αξίζει τον κόπο να διατεθεί στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τον λόγο έχει ξανά η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. Κάποια από τα σχόλια ήδη εκαλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διευκρινίστηκαν όσον αφορά την ευθύνη. Εδώ αναφερόμαστε σε ένα καλύτερο εργαλείο το οποίο θα πρέπει να δυσκολέψει την διάπραξη απατών κατά πελατών πολιτών ενός άλλου κράτους μέλους. Θέλουμε να εξαλειφθούν οι απάτες, να μην ξεγελιώνται οι πελάτες. Κάποιες εταιρείες βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν θα στείλουν τελικά τα αγαθά τα οποία παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν, διότι θα είναι πολύ δύσκολο να ε, προσφύγει ο πελάτης. Εδώ ε, εξετάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις, κατάσταση κατά την οποία έχει πληρώσει κάποιος για κάποια αγαθά και δεν τα παρέλαβε. Αυτό λοιπόν το μέσο, αυτό το εργαλείο μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και στους αγοραστές και στους πολιτές και να θέσει τέρμα στην πολύ κακή αυτή συνήθεια και πρακτική. Αναφερόμενοι σε αυτόν τον κανονισμό δεν μπορώ να παρουσιάσω όλες τις λεπτομέρειες. Θα ήθελα όμως να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους να τους παροτρύνω να διαβάσουν το έγγραφο και να δουν οι ίδιοι πόσο καλό εργαλείο έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ προχωρημένο τεχνολογικά και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παρέμβουμε στον τρόπο λειτουργίας του έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι καλό μέσο, προτείνω κάποιες αλλαγές, κάποιες μικρολεπτομέρειες καλύπτω και νομίζω θα λειτουργήσει άριστα. Η... βάση της πρότασης έχει εξεταστεί ε, διεξοδικά. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέλφους να διαβάσουν προσεκτικά, πολύ προσεκτικά την πρόταση και μετά να προτείνετε τις δικές σας ε, τροπολογίες. Πιστεύω ότι λόγω ελήψεως χρόνου και επειδή η τελική προεδρία ε, είναι πολύ δραστήρια στην όλη προσπάθεια για το θέμα αυτό, για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να τηρήσουμε και εμείς τις προθεσμίες. 27 δηλαδή Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολόγιων και ελπίζω ότι αρχές Δεκεμβρίου θα έχουμε και τη θέση του Συμβουλίου και ελπίζουμε να είναι πολύ κοντά η θέση του Συμβουλίου στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο και μπορούμε να πάμε στο σημείο υπαριθμών 12 όπου θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και συγκεκριμένα στον κύριο Βίκτορ Σολοβέιτσικ ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση για τις διαδικασίες κωδικοποίησης και αναδιατύπωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή να σας δώσω μια σύντομη εξήγηση για τις νομοθετικές τεχνικές της κωδικοποίησης και της αναδιατύπωσης. Όπως ξέρετε, η ενωσιακή νομοθεσία τροποποιείται πολύ συχνά. Μερικές φορές, μετά από την σώρευση τροποποίησεων, μπορεί να οδηγήσει σε κείμενα τα οποία είναι λιγότερο αναγνώσιμα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτές τις τεχνικές της κωδικοποίησης και της αναδιατύπωσης για να απλοποιήσουμε τα νομικά κείμενα και να τα κάνουμε πιο προσβάσιμα και διαφανή. Οι ικανότητες για αυτές τις τεχνικές αναφέρονται σε δύο συγκεκριμένες διαθεσμικές συμφωνίες του 1994 και του 2001. Τι είναι η κωδικοποίηση είναι η διαδικασία για να αντικαταστήσουμε με ένα ενιαίο νομοθέτημα μια υφιστάμενη σε εφαρμογή νομική πράξη που έχει τροποποιηθεί μία ή περισσότερες φορές. Κωδικοποίηση δεν σημαίνει ουσιαστικές αλλαγές στο κείμενο. Οι πράξεις οι οποίες έχουν τύχη κωδικοποίησης ακυρώνονται. Το ουσιαστικό στοιχείο κάθε κωδικοποίησης είναι ακριβώς η απουσία ουσιαστικών αλλαγών. Γι' αυτό οι πραξεις οι οποιες εχουν τυχει κωδικοποιησης ακυρωνονται το ουσιαστικο στοιχειο καθε κωδικοποιησης γίνονται διατηρώντας σταθερή την ισχύ του δικαίου. Και μπορούν να είναι αποδεκτές μόνο αν δεν αλλάζουν την φύση του κειμένου. Αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να πιστοποιηθεί από μια συμβουλευτική ομάδα που περιλαμβάνει εκπροσώπους από την ε, νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν που εξετάζει τις προτάσεις αυτές και επιβεβαιώνει ότι πράγματι πρόκειται μονάχα για δικοδικοποίηση. Η διαδικασία αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να σεβαστούν το γεγονός ότι δεν μπορούν να επιφερθούν ουσιαστικές αλλαγές στην νομοθεσία. Η αναδιατύπωση τώρα είναι μια διαφορετική τεχνική, η οποία συνδυάζει και την κωδικοποίηση και τις τροποποίησεις. Όταν υπάρχει μια αναδιατύπωση υπάρχουν τρεις παρεμβάσεις στο νομοθέτημα. Πρώτα απ' όλα, εισάγονται ουσιαστικές τροπολογίες στο αρχικό κείμενο. Δεύτερον, κωδικοποίηση των μη τροποποιημένων διατάξεων χάρη σε αυτές τις νέες τροπολογίες. Και τρίτον, η ακύρωση του προηγουμένου νομοθετήματος και αντικατάστασή του με το νέο. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι νέες ουσιαστικές διατάξεις και οι αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει να, να εντοπίζονται και να διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες με τη χρήση θεών στοιχείων. Επίσης, και εκεί εμπλέκεται η συμβουλευτική ομάδα των τριών νομικών υπηρεσιών που εξασφαλίζει ότι το κείμενο της Κομισιόν δεν περιλαμβάνει άλλες ουσιαστικές αλλαγές πέραν αυτών οι οποίες έχουν εντοπιστεί και θεοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει πάλι σεβασμός με την φυσιολογική νομοθετική διαδικασία, αλλά θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούν και με το πνεύμα και το γράμμα της διαθεσμικής συμφωνίας και να περιορίζεται η συζήτηση μόνο στα τμήματα της πρότασης που έχουν ταυτοποιηθεί ως νέα στοιχεία. Εάν κατά τη διάρκεια μιας νομοθετικής διαδικασίας φανεί ότι πρέπει να εισαχθούν και άλλες ουσιαστικές τροποποίησεις, ε, πέραν αυτών που έχουν εντοπιστεί, τότε η διαθεσμική συμφωνία σημαίνει ότι αυτές οι πρόσθετες τροπολογίες θα πρέπει πρώτα να, εφαρμοστούν, να προταθούν ε, βάσει των κανόνων που εξασφαλίζουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Επομένως δεν μπορούν στη μέση της διαδικασίας να εμφανιστούν αυτές οι προτάσεις, αλλά απαιτούν μία τροποποιημένη πρόταση από την Κομισιόν για την αναδιατύπωση. Η αναδιατύπωση εξαρτάται από το σεβασμό των κανόνων από όλου του εμπλεκομένου. Στο παρελθόν η Κομισιόν έχει τονίσει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει πιο συχνά τη διαδικασία recast αναδιατύπωση, όπω έχει ζητηθεί και από το Κοινοβούλιο. Αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα, διότι δεν υπήρξε σεβασμό των κανόνων του παιχνιδιού σε μία σειρά από νομοθετικέ διαδικασίε. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν θέλει να επιτύχει το στόχο αυτό και θα περίμενε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμβάλλουν πλήρως για να υπάρξει η πλήρης εφαρμογή του, των κανόνων του παιχνιδιού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο συχνή και αποτελεσματική χρήση αυτής της διαδικασίας της αναδιατύπωσης και είναι στόχος της Κομισιόν να πείσει όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάγκη να χρησιμοποιείται συχνότερα αυτή η διαδικασία. Τέλος, για τις προτάσεις κωδικοποίησης και αναδιατύπωσης που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στη μέση διάταξη της συνεδρίασή σας θα ήθελα να σας πω ότι μετά από το πρόγραμμα κωδικοποίησης του 2008-2009 η Κομισιόν έχει συνεχίσει τις κωδικοποίησεις επί τη βάση ετήσιου σχεδιασμού. Μετά από τη θέση εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν αδύνατο να υπάρξει κωδικοποίηση των νομοθετικών πράξεων, γιατί οι περισσότερε από αυτέ τι πράξει περιλάμβαναν διατάξει επιτροπολογία που έπρεπε πρώτα να ευθυγραμμιστούν με το νέο σύστημα των κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Η έγκριση των τροπολογιών λοιπόν για να γίνει η ευθυγράμμιση με το νέο αυτό σύστημα έδωσε δυνατότητα και πάλι να κωδικοποιούνται οι διάφορες πράξεις. Και έτσι λοιπόν έχετε τις σημερινές προτάσεις για κωδικοποίηση και αναδιατύπωση. Ευχαριστώ. I Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρέγναρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την Κομισιόν τις εξηγήσει αυτές. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα γιατί είχα μια πρακτική εμπειρία με την ε, οδηγία Βρυξέλλες 1 και ε, η οποία υφίστατο τη διαδικασία της αναδιατύπωσης. Η διαθεσμική συμφωνία έχει σαν στόχο να είναι το πλαίσιο για αυτές τις διαδικασίες. Τώρα έχουμε περισσότερες διαδικασίες τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά υπάρχουν πολλές φορές πολλές τροποποιήσεις και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο όγκο τροποποιήσεων και η Κομισιόν θέτει όλες αυτές τις τροπολογίες και εμείς θα ως Ευρωβουλευτές να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το μεγάλο όγκο τροποποιήσεων που δεν είναι εύκολος να τον καταλάβει κανείς. Στην περίπτωση της των, της Βρυξέλλες 1 του, της οδηγίας αυτής, εγώ ενοχλήθηκα γιατί υπήρχε μια πρόταση η οποία δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενεπλέκετο στις περιπτώσεις όπου, πρέπει να υπάρχει, όπου υπάρχει συχνή τροποποίηση, αλλά ήταν μια περίπτωση που ήθελε η Κομισιόν να καταργήσει τη διαδικασία του εκτελεστού τίτλου και ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτήν την ε, ευκαιρία για να τροποποιήσει με αυτόν τον τρόπο αυτή την οδηγία. Και η Κομισιόν τελικά άφησε ελάχιστο χώρο για να αντιμετωπιστούν θέματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, τα οποία είχαν πολιτική σημασία και ουσιαστικά δεν επέτρεψε τη συζήτηση τροπολογιών αυτού του είδους. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και πάλι αυτή τη μέθοδο της αναδιατύπωσης και να εξασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν δεν χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία για να περιορίσει υπερβολικά τους νομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο, και να χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτή τη μέθοδο για να αποκλείσει ορισμένους τομείς όπου πρέπει οι νομοθέτες να αποφασίσουν. Για μένα λοιπόν είναι ουσιαστικό να εξασφαλίσουμε ότι θα ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Για μένα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις, ιδίως για να ξέρουμε ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες μπορούν να υφίστανται κάποια τροποποίηση. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όπως λειτουργεί η διαδικασία περιορίζει τις δυνατότητες του νομοθέτη. Ευχαριστώ. Ζητά κάποιο το λόγο. Δεν θέλει κανείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απαντώντας, να επιβεβαιώσω εκ νέου ότι από την πλευρά μας θεωρούμε σημαντικό για να διατηρηθούν τα δικαιώματα πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα τα θεσμικά όργανα να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την αναδιατύπωση. Για να έχουμε πιο συχνή χρήση της διαδικασίας της αναδιατύπωσης είναι πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες. Ίσως αποδειχθεί αναγκαίο να προσθεθούν κάποιες ε, τροποποίησεις και ίσως τη διαδικασία των συζητήσεων ε, επί του σχεδίου προτάσεως να διαφανεί ότι χρειάζονται και άλλες αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη θα πρέπει να προτείνει τροποποιημένη πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αδίποτε απόπειρα να προσθεθούν ουσιαστικέ αλλαγές στην αδιατύπωση στις διάφορες διατάξεις θα ήταν κάτι που θα υπονόμευε τη βασική αρχή του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς θα παρεμπόδιζε την πιο συχνή χρήση της διαδικασίας αναδιατυπώσεως. Αυτά και ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτού του σημείου. Συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 31. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Νομική Προστασία των Υπηρεσιών που αφορούν ε, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υπό όρους, κωδικοποιημένες υπηρεσίες. Ε, να πω εν είδη εισαγωγής κάποια λόγια. Αυτό το σημείο είναι και το πιο παλιό θέμα που εκρεμεί για την Επιτροπή μας. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπευλήθη το Δεκέμβριο του 2010 εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου. Ανέλαβα εγώ τη συνέχιση του θέματος από τον πρώην πρόεδρο της Νομικής Επιτροπής, από τον κύριο Κάλς Χάινε Λένα. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στην καταπολέμηση των παρανόμων συσκευών που επιτρέπουν την πρόσβαση σε τηλεοπτικές υπηρεσίες χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη πληρωμή και ε, προστατεύουμε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή η προστασία καλύπτει και τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και εκπομπές μέσω του διαδικτύου. Το 1999 το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε τη σύνταξη Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τη νομική προστασία αυτών των υπηρεσιών Πολλές ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ενώσεως μπορούν να αποτελούν παραδείσους για την ανάπτυξη διανομή, κατασκευή συσκευών για την ε, παράνομη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες αν το νομικό ε, πλαίσιο δεν προβλέπει κυρώσεις κατά της συγκεκριμένης δραστηριότητα παραβίασης των συσκευών και των συστημάτων, hacking. Γι' αυτό θεωρήθηκε ότι πρέπει να επεκταθούν οι διατάξει τη οδηγία του 1998 και χρειάζεται ένα κοινό αποτελεσματικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι διαπραγματεύσει που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου τη Ενώσεω υπήρξαν επιτυχεί και η σύμβαση που υιοθετήθηκε το 2001 συνάδει με την οδηγία. Η διατύπωση των δύο κειμένων ε, διαφέρει μόνο σε κάποια σημεία και ελάχιστα. Όμως, πριν ζητήσει το Συμβούλιο από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμβάσεως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διατηνόμενη ότι το Συμβούλιο χρησιμοποίησε λανθασμένη νομική βάση για την απόφαση που αφορούσε την υπογραφή της συμβάσεως. Αντί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εμπορική πολιτική που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο χρησιμοποίησε το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εναρμονίσεως ε, της εσωτερικής αγοράς. Παρόλο που το Κοινοβούλιο δεν έχει ρόλο στη διαδικασία για την υπογραφή της συμβάσεως, αυτή η δικαστική υπόθεση επηρέασε τη δυνατότητα έγκρισης της συνάψεως της συμβάσεως εφόσον το Συμβούλιο έπρεπε να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου πριν ζητήσει την έγκριση από το Κοινοβούλιο. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εξεδόθη τον Οκτώβριο 2013 και στήριξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση. Δικαίω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σωστή νομική βάση, συνεπώ, ήταν το άρθρο 207 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική. Η Ιταλική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλήθησαν να παρουσιάσουν τις εξελίξεις του θέματος και ποια είναι η κατάσταση στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει την πρόταση, πρόκειται να δώσει την έγκριση και περιμένει το σχετικό αίτημα του Συμβουλίου πριν να είναι θέση η Επιτροπή μας να συντάξει ένα σχέδιο εκθέσεως. Να δώσω τώρα το λόγο στον Ζήγα Μπάχοβετς από τη Γενική Διεύθυνση για την επικοινωνία και τα δίκτυα, το περιεχόμενο και τεχνολογία, η DG Connect αυτή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο, κυρία μου, λέει ο πρόεδρος. Ο, συγγνώμη ζητάει ο πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη. Σας αποκάλυψα κυρία μάλλον εννοεί ο πρόεδρος. Με ακούτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι πολύ παλιό θέμα αυτό. Και επειδή είναι παλιό πρέπει να πω ότι από 1η Νοεμβρίου μετακινήθηκε από τη DG Mart στη DG Connect, στη Γενική Διεύθυνση Connect. Είμαστε νέοι όσον αφορά αυτό το θέμα για να συμπληρώσω την ιστορική παρουσίαση του θέματος, τα είπα αυτά. Δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω σε αυτά που εξηγήσατε, Πρόεδρε, διότι πράγματι έχουμε την οδηγία του 1998 ξεκίνησαν έκτοτε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτω ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή και να παρέχεται συγκρίσιμη νομική προστασία και να επιβάλλονται αποτελεσματικές κυρώσεις σε κάποιες χώρες που είναι όμορες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά δεν είναι μέλη αυτής όπως Αλβανία, Σερβία, Ουκρανία, για να παραθέσω κάποιες, όπου υπάρχει μεγάλο εμπόριο, κυκλοφορία αυτών των παρανόμων συσκευών που σπάνε τα συστήματα κωδικοποίησης και υποστασίας. Όπως εξήγησα ήδη, έχουμε πρόταση του Συμβουλίου για την προσχώρηση και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως. Βασιστήκαμε στη διατάξη περισσοτερικής αγοράς της συνθήκης. Το Συμβούλιο θέτησε την προσέγγιση του σε εσφαλμένη νομική βάση Προσεφήγαμε κατά του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όσον αφορά την αποκλειστική αρμοδία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έπρεπε να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείναμε νέα απόφαση του Συμβουλίου για την σύναψη της συμβάσεως για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υπό όρους, conditional access. Αυτό είναι κάτι που συζητείται στις ομάδες εργασίας, μάλλον του Συμβουλίου. Έγινε μια συνεδρίαση νομίζω 3 Νοεμβρίου φέτος στην ομάδα εργασίας για τα οπτικοακουστικά μέσα στο Συμβούλιο. Πρέπει να σταματήσω, διότι η Προεδρία θα πρέπει να σας πει ποια είναι η εξέλιξη του, του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κάρλο Ιμαρίσιο που εκπροσωπεί την Ιταλική Προεδρία. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Εμπρότης να πω ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της συμβάσεως που είναι η καταπολέμηση της πειρατείας που συνδέεται βέβαια στην πρόσβαση πόρους στις υπηρεσίες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα προσχωρεί, συμφωνεί με την ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπό το φως της ε, αποφάσεως του δικαστηρίου η υπόθεση 137 κάθετος 12, 12 και υιοθετήσαμε μετά την απόφαση αυτή το Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο μια νέα απόφαση όσον αφορά την υπογραφή της συμβάσεως αυτή η απόφαση βασιζόταν σε νομικές βάσεις που αποφάσισε το ΔΕΚ. Και αυτή η απόφαση ε, διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση. Αρχές Μαΐου. Το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα. Έγκριση της αποφάσεως για την σύναψη της συμβάσεως. Εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως, η εξέταση του κειμένου στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Προτάθηκαν τροποποίησεις στη Σύμβαση. άθρο για το άρθρο 9 και 10 και δημιουργούν κάποιες αβεβαιότητες. Αυτά τα άρθρα δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πλήρως την αποκλειστική της αρμοδιότητα. Εφόσον βάσει του άρθρου 9 της συμβάσεως, ο αριθμός των ψήφων που Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε στις διαβουλεύσεις πολυμερείς αντιστοιχεί στον αριθμό ψήφων των κρατών μελών που είναι μέρη της συμβάσεως, συμβαλόμενα μέρη. Αυτό συζητείται ακόμα στην ομάδα εργασίας, στο Συμβούλιο. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση. και θα υποβληθεί στο Κορεπέρ. Ελπίζουμε να υποβάλουμε τη λύση αυτή μέχρι το τέλος του έτους, πιθανότατα τον μήνα Δεκέμβριο. Αφού επιτευχθεί αυτό και αφού ολοκληρωθούν τα πάντα, θα υποβληθεί το κείμενο στο Κοινοβούλιο ζητώντας ε, την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Πιστεύει το Συμβούλιο ότι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ενωμική Επιτροπή ε, είναι απαραίτητη για αυτό το θέμα. Πάντα το πιστεύω με αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Σας ευχαριστώ που μας περιγράψατε την όλη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει η συζήτηση, να ακούσουμε τις απόψεις των μελών, υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο το λόγο. Οπότε, επόμενο βήμα είναι το εξής το Συμβούλιο επίσημα θα ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την σύναψη της σύμβασης αυτής και από τη στιγμή που θα ληφθεί αυτή η αίτηση αυτό, εγώ θα πρέπει να συντάξω σχέδιο εκθέσεως που θα συζητηθεί εν συνεχεία στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ, <clears throat> δεν μπορώ επομένως να θεωρήσω λήξαν το θέμα αυτό. Θα προχωρήσω στο 33. ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας για τα εγκληματολογικά και θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας, τον αξιότιμο κύριο Μαρίνιου Ιππίντου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για να μπορέσει η Επιτροπή μας να δώσει μια γνωμοδότηση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αναδιάθεση του Eurojust που αντιμετωπίζεται τώρα στην Επιτροπή των Δημοσίων Ελευθεριών. Θα ήθελα από τώρα να πω ότι το θέμα αυτό έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο μια συζήτησης και μια έκθεση στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Βος ήταν και παρόν τότε και ήταν ο αρμόδιος για μια εργασία η οποία εμένα μου φαίνεται ότι καλύπτει πλήρως τα ουσιώδη θέματα και τα οποία ε, διακυβεύονται σε αυτήν την περίπτωση το να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε το Eurozoo είναι κάτι το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Όπως είπε και ο κύριος Βος, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν ερωτήσεως και για τα οποία πρέπει εμείς να εκφέρουμε γνώμη. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων και σε σχέση με την αρχή η οποία θα είναι αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα συλλεγούν. Στην προηγούμενη έκθεση να το πω καλύτερα. Η Europol, η οποία ήταν στην περίπτωση Europol, η αρχή η οποία εποπτεύει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων. Και εδώ θα πρέπει πιστεύω να έχει τον ίδιο ε, ρόλο για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των ε, διαδικασιών. Επίσης, ποια θα είναι η αλλαγή στο καθεστώς της Eurojust και της Europol. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Φυσικά, προκύπτει όλο αυτό το θέμα λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως της ε, εγκληματικότητας η οποία είναι υπεροργανωμένη σε οικονομικό επίπεδο, διάφορες μορφές λαθρεμπορία, η υπερική πορνογραφία. Η απάντηση λοιπόν στα θέματα αυτά είναι κατά την απόψή μου δύσκολη και έχουμε το εξής πρόβλημα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν, έχει, δεν έχουμε προβεί σε μία ε, κατά κάποιο τρόπο ταξινόμηση σε διάφορες κατηγορίες των αδικημάτων και δεν έχουμε θεσπίσει την έννοια του ομοσπονδιακού εγκλήματος ούτως πίν μια προσβολή στην νομική τάξη της Ένωσης και όχι μόνο των κρατών μελών, <clears throat> αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για την ύπαρξη ενός όργανου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ερευνά αδικήματα, των οποίων, για τα οποία η αρμοδιότητα καταρχήν ανήκει στα κρατή-μέλη. οι εισαγγελικέ αρχές, οι αστυνομίε των κρατών μελών ή οι <clears throat> δικαστικές αρχές όταν έχουν τον ρόλο για, τις, για τα προβλήματα αυτά. Το να δημιουργήσουμε λοιπόν ευρωπαϊκά όργανα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ερευνήσουμε αδικήματα των οποίων η αρμοδιότητα βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των κρατών μελών αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και για τα οποία θα πρέπει να εκφέρουμε γνώμη. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα τα οποία συνάπτονται με την φύση των ε, αξιωματούχων του Eurojust, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, αν θα πρέπει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος να είναι υπάλληλοι της Eurojust ή αν θα πρέπει να είναι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αμείβονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και εγώ με μεγάλη προσοχή θα μελετήσω το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρα στο παρελθόν ο κύριος Αντιπρόεδρος Άξελ Βος, γιατί νομίζω ότι ήδη περιλαμβάνει τα κέρια σημεία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σωστή γνωμοδότηση στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Thank Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Πίντου που αναφέρθηκε και στην έκθεση Eurojust και η σχετική μεταρρύθμιση σχετίζεται και με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής αγγελίας που δεν ξέρουμε βέβαια που θα καταλήξει η προσπάθεια αυτή και αν θα καταλήξει. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να προσαρμόσουμε την Eurojust. Στην έκθεση που είπατε είχαμε παρακαλέσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει τι στάση θα κρατήσει για τη μεταρρύθμιση της Eurojust εφόσον καταλήξει μοναχά σε διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα χρειαστεί βέβαια να περιμένουμε μέχρι ότου γνωρίζουμε τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να κάνουμε και την μεταρρύθμιση της Eurojust. Κατά βάση, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, βρισκόμαστε σε ένα κατόφλιο, να δούμε δηλαδή εάν θα δημιουργήσουμε και ποινικό σκέλος του ευρωπαϊκού δικαίου. Έχουμε την Ευρωπόλ, το αστυνομικό, τον αστυνομικό πόλο, έχουμε το δικαστήριο. Αυτό που δεν έχουμε είναι ένα δικαστήριο, ειδικό, ποινικό δηλαδή, και διαδικασίες. Φαίνεται να λείπει η πολιτική βούληση και το πολιτικό θάρρος. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα δεκαριά δεκαετία-δεκαπέντε χρόνια πριν να τα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Μακάρι να γινόντουσαν από την αρχή σωστά τα πράγματα. Πάντως, σε ό,τι αφορά το ουσιώδε περιεχόμενο τώρα, θα εξετάσουμε την ενδεχόμενη σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ Eurojust και ε, Ευρωπαϊκή Αγγελία, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κιόλα κατά πόσον οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο συλλογικό σώμα αλλά και στο εκτελεστικό όργανο του Eurojust, γιατί άραγε είναι απαραίτητη. Εμένα δεν μου φαίνεται απαραίτητη η παρουσία του εκεί και το ζήτημα της έδρας που βεβαίως σχετίζεται Εφόσον πρόκειται να συνεργαστούν οι δύο αυτοί οργανισμοί θα πρέπει να έχουν κοινή έδρα. Επίσης το δημοσιονομικό ε, ζήτημα. Εγώ θα τα πω αυτά βέβαια και στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Θα προτείνω να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εγγελίας, πώς θα προχωρήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ορθώς και απέναντι στην μεταρρύθμιση Eurojust. Ευχαριστώ Κάφμαν. Η κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ και τους δυο συναδέλφους που μίλησαν. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπαν. Σύμφωνα με το άρθρο 85 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης, ο Γιώργο στην οργανισμό. Και εκεί μπαίνουν και κάποια διαδικαστικά θέματα. Μπαίνει ταυτόχρονα το θέμα και τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι κάνει το Συμβούλιο. Θα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώ έχουν προχωρήσει οι διαβουλεύσει στο Συμβούλιο για το ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τη σχέση μεταξύ Eurojust και Εισαγγελίας. αν εξετάσει κανείς τις πηγές, τα κείμενα δηλαδή, θα δει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δραστηριοποιείται μόνο εφόσον πρόκειται για ποινικά αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ορισμός είναι ξεκάθαρος. Στο Eurojust όμως υπάρχει και το παράρτημα 1, όπου διαλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Άρα είναι κέρια σημασία θέμα. Δεν ξέρω τώρα το Συμβούλιο αν έχει στο μεταξύ πει κάτι σχετικά και έχει διαλύσει τα νέφη. Τώρα επανέρχομαι σε κάτι που είπε ο Μαρίνιου Ντεπίντου, τη σχέση δηλαδή με την Ευρωπόλ. Και εδώ σημειώνεται ένα πρόβλημα. Αν δείτε την λίστα των ε, αδικημάτων, είναι διαφορετική η λίστα στην Ευρωπόλ και διαφορετική εδώ. Δεν είναι δυνατόν αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν. Τελευταία δε παρατήρηση έχει ως εξής. Για την πρόταση για την Eurojust, στην πρόταση μόνο για την Eurojust, λέγει ακόμη ότι οι εθνικές βουλές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την διαχείριση της Eurojust. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να το θέσουμε υπόψη και των εθνικών βουλευτών, διότι πρόκειται για γενικό θέμα. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, και ο Eurojust θα είναι ο οργανισμός, χρειάζονται κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτό πρέπει να ισχύει και για άλλους οργανισμούς, από τους οποίους έχουμε πληθώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ μονάχα σε δύο σημεία για αυτά που ελέγχθηκαν για την προηγούμενη ομιλήτρια. Η σχέση Europol και Eurojust ως νομομαθής με ανθρωπιστική παιδεία και ανοιχτό στα θέματα του κράτους δικαίου, πιστεύω ότι πάντα η αστυνομία πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των εισαγγελικών αρχών στη δική μου χώρα γίνεται έτσι. Πάντα πρέπει να υπάρχει εποπτεία της αστυνομίας από τους εισαγγελείς. Υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις χώρες και στη δική μου χώρα υπάρχουν πάντα σχέσεις μεταξύ των δικαστικών και της αστυνομίας. Η αστυνομία βάσει του νόμου εξαρτάται η αστυνομία η οποία είναι αρμόδια για τις ε, ανακρίσεις εξαρτάται κατευθείαν από την κυβέρνηση μέσω των εισαγγελικών αρχών αλλά ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός προέρχεται από το, την κυβέρνηση όλα τα απαραίτητα γίνονται σε διοικητικό επίπεδο από την κυβέρνηση αλλά δεν έχει διοικητική εξάρτηση από το, τις εισαγγελικές αρχές. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε αμφιβολίες και δυσκολίες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται ορισμένες ε, ε ανακρίσεις και σε προβλήματα και αποτυχίες για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το θέμα λοιπόν της ε, εξόχως οργανωμένης εγκληματικότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αγώνας λοιπόν κατά της εγκληματικότητας είναι μια απέτηση των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Όταν έχουμε μια χώρα, όταν έχουμε ένα έδαφος, όταν δεν τηρείται η νομοθεσία και όπου δυσκολεύονται οι δικαστικές έρευνες, αυτό είναι ένα κίνητρο για την εγκληματικότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητε της με όλα τα κακά που συνεπάγεται αυτό για την κοινωνία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Μπορούμε να κλείσουμε προς το παρόν το σημείο αυτό και να περάσουμε στο σημείο 34, στο οποίο αφορά την πρόταση να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστικών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πάλι ο κύριος Μαρίνιου αλλά και Πίντου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για μια έκθεση στην οποία εγώ έχω αναλάβει την εισηγεσία. Αυτή πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη, για την τροποποίηση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο. Η δικαστική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όπως ξέρετε η εξής. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πιο κάτω έχουμε το, το Πρωτοδικείο και επίσης το Δικαστήριο για την Δημόσια Διοίκηση για τους ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο έχει ήδη παρουσιάσει εδώ και τέσσερα χρόνια μια πρόταση για να αυξηθεί ο αριθμός των πρωτοδικών από 28 σε 40. Αυτή η πρόταση ενεκρίθη και το πρόβλημα προέκυψε μονάχα όταν είχαμε να προχωρήσουμε στον διορισμό των δικαστών, το πρόσθετο των δικαστών, διότι τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Τα κράτη-μέλη είναι 28. που είναι ο τωρινός αριθμός των ε, μελών του πρωτοδικείου. Εάν αυξηθεί όμως ο αριθμός των δικαστών και φτάσει στους 40, θα χρειαστεί να διορίσουμε 12 πρόσθετους δικαστές, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη για το ποιος θα προέλθει από πού, εφόσον είναι μικρότερο αριθμό από τον αριθμό των κρατών μέλων. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση εμπλοκή και αδιεξόδου που έχει επανέλθει στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενδιαμέσω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προτείνει μια νέα τροποποίηση. Δηλαδή, αντί να αυξηθεί μονάχα ο αριθμό των κρατων μελων υπαρχει λοιπον μια κατασταση εμπλοκη και αδιεξοδου που εχει επανελθει στα χερια του ευρωπαικου κοινοβουλιου αμέσως κατά 12, να προσθεθούν 28 δικα... πρόσθετοι δικαστές να φτάσουμε σε 58 ε, δικαστές, να μην έχουμε πια ένα πρωτοδικείο και ένα δικαστήριο για τη δημόσια διοίκηση, να έχουμε ένα κοινό δικαστήριο το οποίο θα καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο όμως χάνεται ένας βαθμός δικαιοσύνης και περνάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να έχει 56 δικαστές, αλλά να μην υπάρχει πρωτοδικείο ή δικαστήριο για τη δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε εξετάσει σε μια συνάντηση που προέδρευσε ο Πάβελ Σβόμποντα όταν ήταν παρόντες οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και μας παρουσίασαν την επιχειρηματολογία για την αλλαγή αυτή, όπως ε, αναφέρθηκε ήδη από τον πρόεδρο στην αρχή της συνεδρίασης. Θα πάμε και στο ακριτικό Λουξεμβούργο στις 3 Δεκεμβρίου. Στρασβούργο λέει ο, ο στο Λουξεμβούργο διορθώνει για να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση και να έρθουμε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να μπορέσουμε να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες επιτοπίως και στη συνέχεια να εκμεταλλευτούμε αυτές τις πληροφορίες που θα έχουμε συλλέξει, ώστε να παρουσιάσουμε μία πρόταση για τροποποίηση. Το κέριο θέμα, το κεντρικό θέμα τώρα είναι το εξής. Υπάρχουν εκατοντάδες διαδικασιών εν εξελίξη που έχουν εκδοθεί ο αριθμός των αποφάσεων που έχουν ληφθεί είναι πολύ μικρότερος από των διαδικασιών που εκκρεμούν. Το θέμα είναι αυτές οι διαδικασίες που εκκρεμούν, που είναι να εξελίξει Ποιος είναι ο πιο απλός, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο λιγότερο πολυδάπανος τρόπος για να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις. <clears throat> και το θέμα είναι μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα άλλο τρόπο να αυξήσουμε όχι τους δικαστές αλλά το τεχνικό προσωπικό, τους ε, εισηγητές ή τους <clears throat> συνεργάτες των δικαστών. Υπάρχει λοιπόν μια γενική προβληματική για να δούμε ποιος είναι ο λιγότερο πολυδάπανος τρόπος για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι μπορούμε, όπως είπε και συγητής, να πούμε ότι η κατάσταση στο ΔΕΚ έγινε αφόρητη. Πάνω από τρία χρόνια όλος ο κόσμος συμφωνεί. Πράγματι πρέπει να αυξηθεί ο των δικαστών του πρωτοδικίου και έχουν σωρευτεί καθυστερήσεις παρά τις διάφορες τροποποίησεις που έκανε το δικαστήριο όσον αφορά τη μέθοδο Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και για ένα κράτος δικαίου αυτό είναι απαράδεκτο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι πολύ αργή. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών. Πρέπει να πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι η πρόταση για διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών του πρωτοδικίου θεωρούσε ότι ήταν υπερβολικό σαν πρόταση. Υπάρχει συμφωνία ότι χρειάζονται παραπάνω 9 με 12 δικαστές και πάντα θεωρούσα ότι θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα κυκλικής αναλλαγής, ούτω ώστε να διορίζονται οι δικαστές που πρέπει. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τους δικαστές στο Λουξεμβούργο, αλλά νομίζω ότι το μπαλάκι είναι στην πλευρά του Συμβουλίου θετική άποψη του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε κάποια συνένεση. Θα πρέπει λοιπόν να ανεχθούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Και θα πρέπει να κινηθούμε προς όφελος του δικαστηρίου και των Ευρωπαίων πολιτών που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κυρία Ντίεφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, έχουμε όλοι λάβει την επιστολή που απεστάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον κύριο Σκούρη στις 13 Οκτωβρίου. Να υπογραμμίσουμε την περίπτωση που αναφέρεται στην επιστολή και αφορά και το θέμα που συζητούμε. Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το δικαστήριο όσον αφορά το διορισμό ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Δημόσιας ε, Δίκησης. Λοιπόν, το δικαστήριο έχει μόνο 7 δίκαστες, διορίζονται από το Συμβούλιο, ομόφωνα, μετά από μια διαδικασία επιλογής που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει καταλόγου υποψηφίων που καταρτίζεται από μια εξάρτητη επιτροπή. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 η θητεία δύο μελών του δικαστηρίου εξέπνευσε και το Συμβούλιο πρέπει να ακολουθεί στη διαδικασία το διορισμό δύο νέων δικαστών. Αυτό δεν έγινε. Έτσι δε περαιτέρω η Προεδρία του Συμβουλίου φαίνεται να πιστεύει ότι η διαδικασία διορισμού θα πρέπει να ανασταλεί αναμένοντας απόφαση για μια συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βάσης μεταρρύθμισης αυτής το Δικαστήριο της Δημοσίας Υπηρεσίας και το Γενικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγχωνευτούν τον Οκτώβριο του 2016. Ακόμα και αν εγκριθεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αυτή η πρόταση, η εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το 2016. Μέχρι τώρα έχουν διοριστεί τρεις υποψήφοι. Ο παρόν πρόεδρος του δικαστηρίου και άλλοι δύο υποψήφοι από τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία ο Βούλγαρο και ο Πορτογάλο υποψήφιο την χάνουν υποστήριξη τη πλειοψηφία των κρατών μελών. Ο διορισμός του όμω έχει ανασταλεί από το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα η θητεία δύο μελών του δικαστηρίου έχει εκπνεύσει. Έχει λήξει. Πρόεδρε, πιστεύω ότι η αναστολή αυτή οδηγεί σε έλλειψη ασφαλείας δικαίου, παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου και προφανώς είναι εις βάρος της σωστής απόδοσης της δικαιοσύνης. Έτσι δεν περαιτέρω. Αν δεν διοριστούν αυτοί οι δύο νέοι δικαστές, με το μη διορισμό των δύο νέων δικαστών, το Συμβούλιο δεν συμμορφώνεται με τι υποχρεώσει που απορρέουν τη συνθήκη. Ο πρόεδρο Κουρή ο ίδιο είπε ότι ήδη είμαστε μάρτυρες των αρνητικών συνεπειών του αδιεξόδου. Επηρεάζεται η ορθή απόδοση του δικαιοσύνη διότι η έλλειψη ασφαλείας δικαίου δεν επιτρέπει την ορθή διαχείριση, εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων. Εάν υπάρχει εκπρόσωπος του Συμβουλίου, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί η διαδικασία διορισμού μελών του Δικαστηρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας έχει ανασταλεί και γιατί εξαρτάται από τη μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου. Γιατί ζητήθηκε από το Συμβούλιο να ανενώσει τη θητεία των δύο μελών του Δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου του τότε πρόεδρου του κ. Πολ Μαχώνη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και παρόλα αυτά το Συμβούλιο αρνήθηκε να το κάνει αυτό και διόρισε δύο υποψηφίους από τον κατάλογο βάσει της ε, ε, κυκλικής εναλλαγής. Δεν πιστεύετε ότι το πάγωμα της διαδικασίας διορισμού δημιουργεί ανησυχίες περί διακρίσεων και περισσότιμου αντιμετωπίσεως, διότι παρόμοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα η Επιτροπή μας θα μπορεί να θέσει προφορική ερώτηση επ' αυτού στο Συμβούλιο. Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε εμείς να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του δικαστηρίου, ενώ επιδεινώνται τα προβλήματα από το Συμβούλιο. Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, με τα χαράς να σας τις δώσω. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει παρόν εκπρόσωπος του Συμβουλίου για να μπορέσει να απαντήσει. Ίσως μπορεί ωστόσο αργότερα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Λεμπρετών. On a évoqué Ακούστηκε πριν για εθνικές γραφειοκρατίες. Ωστόσο, ποτέ δεν αντιδρά κανείς όταν πρόκειται για αύξηση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί. Και τώρα το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πλήττεται από το ίδιο φαινόμενο, διότι μας προτείνουν εντελώς παράλογα να διπλασιάσουν τον αριθμό των δικαστών, περνώντας από 28 σε 56. Εγώ προσωπικά βλέπω εδώ δύο ενστάσεις. Πρώτη, οικονομική. Διότι θα αυξήσει κι άλλο το κόστος της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης. Διάφορες έρευνες έχουν καταλήξει ότι ένας δικαστής κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Άρα εδώ θα έχουμε άλλα 28 εκατομμύρια τον χρόνο. Και σας υπενθυμίζω ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό αντιμετωπίζει σοβαρότατα ελλείμματα. Ήδη κατά παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει εδώ μέσα να γίνουμε λογικοί. Σηκώνουμε το δάχτυλο για να μαλώνουμε τις χώρες μέλη, αλλά όχι τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα. Το άλλο είναι πολιτικό το σχόλιο. Αυξάνοντας τόσο σημαντικά τον αριθμό των δικαστών, θα δώσουμε πολύ μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη από αυτήν που έχει. Είναι λοιπόν αυτό επιθυμητό από την άποψη της δημοκρατίας. Το δικαστήριο αυτό θα έχει τόσο ελεύθερο χρόνο που για να αυτοαπασχοληθεί προτείνει να περιλάβει και το πρωτοδικείο δημόσιας διοίκησης. Και δεν φτάνει και αυτό. Γνωρίζουν όλοι ότι ένα όργανο εφόσον υπάρχει δημιουργεί και απασχόληση για τον εαυτό του. Πώς θα απασχοληθούν αυτοί οι δικαστές αναπτύσσοντας όλο και περισσότερο αρχές που ξεφεύγουν από τις συνθήκες. Το, η αρχή της ε, του ε, πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι κάτι που είναι αυτονόητο, το έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τον φόρτο εργασία του δικαστηρίου. Ας εμπνευστούμε από το γαλλικό μοντέλο με πολύ πιο σύντομες αποφάσεις. Άλλο θα μπορούσε να είναι να εμπνευστούμε από το αμερικανικό μοντέλο με ένα ανώτατο δικαστήριο που το οποίο θα επιλέγει τις, τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του. Κύριος Βούδας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες ε, σκέψεις για το θέμα αυτό και μόνο. Ελέγχθη ότι ένα δικαστήριο δεν μπορεί πια να αντιμετωπίσει το, το φόρτο εργασίας του. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Με το να διπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών σε 56 δεν λύνουμε τα προβλήματα επειδή ήδη κοστίζει ένα εκατομμύριο το χρόνο ο κάθε δικαστής. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε ένα σύστημα εκπεριτροπής ώστε οι δικαστές οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον να δίδονται από τα κάτι μέλη με βάση εκπεριτροπής διορισμού. Δεν είναι λύση μόνο να προκρίνουμε τη λύση του διπλασιασμού των αριθμών των δικαστών για να λύσουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε και τις διαδικασίες γιατί αν όταν η δικαιοσύνη αποδίδεται καθυστερημένα είναι σαν να μην υπάρχει δικαιοσύνη. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Μήπως το Συμβούλιο θέλει να πει κάτι. Merci, ευχαριστώ. Η Προεδρία του Συμβουλίου δεν είναι παρούσα, αλλά ως νομική υπηρεσία του Συμβουλίου δεν μπορώ να εκφράσω την πολιτική θέση του Συμβουλίου, απλώς θέλω να θίξω ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με την παρατήρηση που έγινε για το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Δεν υπάρχει καμία απόφαση να καταργηθεί αυτό το δικαστήριο όπως ελέγχθη. Απλώς υπάρχει ένα μπλοκάρισμα γιατί χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Από τη που δεν υπάρχει ομοφωνία για τον διορισμό, για την κάλυψη δύο θέσεων οι οποίες θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί το Σεπτέμβριο του 2014, εφόσον δεν υπάρχει λοιπόν συμφωνία για να διοριστούν οι δύο αυτοί δικαστές στο Δικαστήριο Δημόσιας όπου χρειάζεται ομοφωνία, η κατάσταση είναι μπλοκαρισμένη. Δεν φταίει κανεί, απλώ δεν έχουμε βρει την ομοφωνία, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν λιγότερα μέλη αυτού του δικαστηρίου από ότι κράτη-μέλη που εκπρόσω που παίρνουν την απόφαση. Δόθηκε ένας κατάλογος έξι ονομάτων για τις δύο αυτές θέσεις, μεταξύ των οποίων και ο τωρινός πρόεδρος, ένας Πορτογάλος υποψήφιος, ένας Βούλγαρος υποψήφιος στην τρίτη θέση, και άλλες εθνικότητες και υπάρχουν μόνο δύο θέσεις. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια πολιτική συμφωνία για να καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν μέχρι στιγμής και μάλλον βραχυπρόθεσμα θα είναι αδύνατο να βρεθεί μια συμφωνία. Γι' αυτό η Προεδρία του Συμβουλίου πρότεινε στο δικαστήριο να κάνει νέες προτάσεις και το δικαστήριο ήρθε με την πρόταση αυτή την συνολική που θα την εξετάσετε και στο μέλλον σίγουρα που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα αν υποστηριχθεί από το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο γιατί έτσι λύνεται το θέμα και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου για τη Δημόσια Διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα της εμπλοκής και θα μπορέσουν έτσι με τον τρόπο αυτό να διοριστούν πολύ γρήγορα οι δύο δικαστές μέχρι ότου απορροφηθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ένας από τους ε, καλεσμένους, ο κύριος Κάρλος Εσκομπάρ, γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ίσως μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί πρόκειται για τη λειτουργία αυτού του οργάνου απόδοσης δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα γέννη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις επιχειρήσει και για τους απλούς πολίτες. Νομίζω πολύ σωστά το έχει υπενθυμίσει ο εισηγητή σα το ιστορικό της πρόταση του δικαστηρίου, γιατί υπήρχαν τρία χωριστά δικαστήρια. Το δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τις οικονομικές διαφορές για τα μέτρα περιοριστικά που αναλαμβάνει το Συμβούλιο εναντίον ορισμένων ατόμων, αλλά εδώ και χρόνια αυτό το δικαστήριο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην αύξηση του όγκου εργασίας του. Γι' αυτό το δικαστήριο είχε προτείνει να υπάρξει μια αύξηση κατά 12 του αριθμού των δικαστών του. Υπήρξε συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά και υπήρξε κάποια συμφωνία σε επίπεδο συμφωνίου παρά το γεγονός ότι το θέμα της κατανομής αυτών των 12 προσθέτων θέσεων, που είναι λιγότεροι βέβαια τα κρατημέλη, παρέμεινε. Υπήρξε λοιπόν η αίτηση της Ιταλικής Προεδρίας να υποβάλει νέες προτάσεις στο δικαστήριο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να δούμε αν <clears throat> σε σχέση με την κατάσταση η οποία λειτουργούσε το 2011 τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή αν έχουν επιδεινωθεί. Για μας αυτό το σημαντικό είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την τροποποίηση της κατάστασης. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ακόμα σημαντικότερη αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε το 2011. Το τέλος, στο τέλος του 2010 είχαμε 636 υποθέσεις. Εφέτος προβλέπεται να έχουμε 950 υποθέσεις μέσα σε τέσσερα χρόνια μια αύξηση περίπου 50%. Και αυτή είναι μια πιο γρήγορη αύξηση από ό,τι περιμέναμε. Εμείς μπορεί να ε, θεωρούσαμε ότι θέλουμε 5 ή 6 δικαστές παραπάνω, αλλά αυτό τώρα πρέπει να προσαρμοστεί στον αριθμό των υποθέσεων που έρχονται ενώπιόν μας. Υπάρχει ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων που ήταν 1.300, τώρα στο τέλος του χρόνου θα είναι πάνω από 1.500. Υπάρχει λοιπόν η μη ικανότητα του δικαστηρίου να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσα σε λογικά χρονικά διαστήματα. Είναι το θέμα λοιπόν του χρόνου εκδίκασης που είναι το άλλο στοιχείο που είχε υπόψη το δικαστήριο όταν έκανε αυτή την πρόταση. Από το 2011, 8 φορές διεπίστωσε το δικαστήριο ότι διαδικασία είχε ξεπεράσει το άρθρο 47 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δηλαδή το δικαίωμα να υπάρξει μια λογική διάρκεια της διαδικασίας. Υπήρξαν τέσσερις προσφυγές ήδη <clears throat> επί τη βάση αυτής της διαπίστωσης που υπευλήθησαν από ευρωπαϊκές εταιρείες ζητώντας αποζημίωση λόγω του υπερβολικού μήκους της διαδικασίας που παραβιάζει το άρθρο 47. Το συνολικό ποσό που έχει αιτηθεί από αυτές τις εταιρείες ξεπερνάει τα 23 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Να, τα οικονομικά στοιχεία. 23 εκατομμύρια ευρώ για επανόρθωση ζημιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαδικασίες, τέσσερις διαδικασίες <clears throat> όπου οι ετούντες θεωρούν ότι ήταν υπερβολική η διάρκεια της διαδικασίας. Η ανάλυση λοιπόν του δικαστηρίου είναι ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, έχει επιδεινωθεί προς το χειρότερο από ό,τι περιμέναμε το 2011. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους για να ανταποκριθούμε <clears throat> στην αίτηση της Προεδρίας του Συμβουλίου και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αποφεύγων συγχρόνως τα πολιτικά προβλήματα τα οποία έχουν τροχοπεδίσει στη διαδικασία. Γι' αυτό έχετε ενώπιον σας αυτή την πρόταση επειδή φυσικά εσείς θα έχετε την ευκαιρία να το συζητήσετε και με τους ε, δικαστές όταν έρθετε στο Λουξεμβούργο θέλω να σας αναφέρω περί τίνος πρόκειται και να διευκρινίσω ορισμένα στοιχεία. Καταρχήν δεν διπλασιάσουμε τα δικαστήρια. Είχε προταθεί να έχουμε 12 ε, δικαστές <clears throat> από τους οποίους 7 οι δικαστές του Δικαστηρίου Δημοσίας Δίκησης υπάρχουν ήδη το 2009 προσθέθηκαν ε, ναι, νέα πρόσθετοι δικαστές και ο, ο στόχος της πρότασης είναι να έχουμε ένα δικαστήριο το οποίο θα είναι το πρωτοδικείο και ένα το οποίο θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με διπλάσιο αριθμό μελών. Έτσι ξεπερνούμε το πολιτικό πρόβλημα <clears throat> και κάνουμε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του όγκου εργασίας. Να πω κάτι για το κόστος. Μιλήσατε για ένα εκατομμύριο αναδικαστή. Το κόστος στην πρώτη φάση, οι 12 δικαστές που ζητήσαμε από το 2011, είναι 11,6 εκατομμύρια αναφέρεται στο έγγραφο, αλλά είναι 9,8 στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε τους φόρους και όλα αυτά. 9,8 μαζί με το κόστος υποδομής, το κόστος της γραμματιακής υποστήριξης 9,4 όχι 9,8 για τη δεύτερη δόση που είναι οι 7 δικαστές του πρωτοδικίου ε, δημόσιας διοίκησης είναι 1,7 δισεκατομμύρια και για την τρίτη φάση από το 2019 για τους τελευταίους 9 δικαστές θα είναι 7,2 εκατομμύρια. Δηλαδή για τους 28 δικαστές το συνολικό κόστος θα είναι 18,5 εκατομμύρια. Που είναι πολλά λεφτά, αλλά είναι 6,6% του προϋπολογισμού του δικαστηρίου. Δεν εκρήγνεται ο προϋπολογισμός του δικαστηρίου και 0,3% του συνολικού διοικητικού προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών οργάνων. Και αυτό είναι το κόστος του να εξασφαλίσουμε ότι η δικαιοσύνη στην Ευρώπη θα λειτουργήσει σωστά. Και ένα τελευταίο στοιχείο και κλείνω. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε το κόστος της μη μεταρρύθμισης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν <clears throat> αγωγές για αποζημίωση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες που είναι εκκρεμής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που και αυτές επέχουν τον κίνδυνο μιας τέτοιας προσφύγης ενώπιον του δικαστηρίου για καθυστέρηση. Δεν λέω θα κερδίσει αυτός ο οποίος κάνει την αγωγή, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος. Και επίσης το κόστος της ε, διαδικασίας. Έχουμε καταρχήν διαδικασίες ακύρωσης των προστήμων που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού. Οι λογιστές της Κομισιόν στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 αποτίμησαν αυτές τις, αυτά τα πρόστιμα συνολικά σε 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μπλοκαρισμένα σε λογαριασμούς περιμένοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα χρήματα αυτά δεν είναι στα χέρια των επιχειρήσεων που προσφεύγουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουν λοιπόν τα ποσά αυτά ούτε μπορούν να μπουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο δεν υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Και επίσης υπάρχουν οι διαδικασίες για κρατικές επιδοτήσεις που είναι ακόμα πιο μεγάλα ποσά που ξεπερνούν λοιπόν κατά παρασάγκα στο ύψος των προστήμων. Σχέση κόστους-οφέλους. Από οικονομική άποψη για μας είναι απόλυτα λογικό <clears throat> για λιγότερο από 20 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσουμε στην τελική αυτή φάση το 2019 σε ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και αυτό πρέπει να το συγκρίνουμε με τα πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά επίση υπάρχει και η αξία τη καλή λειτουργία τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και η αξία του σεβασμού του κράτου δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο σα έχουμε υποβάλει αυτή την πρόταση, αναμένων ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω έχει κάνει μέχρι τώρα, θα υποστηρίξει το δικαστήριο στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σάντρουσον. Ενδιαφέρον που ακούσαμε ότι αυξήθηκε η δηλαδή ο αριθμός των υποθέσεων και τόσο πολύ μάλιστα. Διερωτώ με τώρα. Ο κύριος Κάρλο Εσκομπάρ Ξέρει την απάντηση. Γιατί αυξήθηκαν τόσο πολύ. Είναι μόνιμη αυτή η αλλαγή. είναι κακή συγκυρία. Θέλετε να απαντήσετε, λέει ο Πρόεδρος. Και ο κομπάρ μάλιστα. Για διαφόρους λόγους αυξήθηκε ο αριθμός των υποθέσεων η αύξηση της νομοθετικής δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσο αυξάνεται η εκπόνηση δικαίου ευρωπαϊκού, υπάρχουν και υποθέσεις που γεννώνται από την εφαρμογή των κανόνων. Και οι εταιρείε ε, κινούνται διασυνοριακά. Υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών και δημιουργούνται οικονομικές διαφορές. Υπάρχουν θέματα τεχνικής φύσεως, ε, θέματα μάρκας ε, ε, μετά την ε, οδηγία REACH για τις χημικές ουσίες από το Ελσίνκι. Υπάρχουν ε, διαφορές για περιοριστικά μέτρα που υιοθετούνται κατά υπηκών τρίτων χωρών στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Ρώσοι, Ουκρανοί, Ιρανοί κλπ. Διάφορα μέτρα και προξενούνται διαφορές υπάρχει ε, καμία εκατοστή τέτοιων υποθέσεων. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση των υποθέσεων και επιμονή μου βάσος. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας είπα ότι προετοιμάζομαι ένα έγγραφο συμπληρωματικό με αυτά τα στοιχεία που σας παρέθεσα που θα σας δείξουν, θα σας στείλουμε το έγγραφο βέβαια, δείχνουν τα στοιχεία λέω πως αυτή η τάση είναι μόνιμη. Δεν είναι συγκυριακή, αλλά είναι σταθερή η τάση αυτή η αυξητική. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Καπένε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν το δικαστήριο ζήτησε καταρχάς την αύξηση αριθμού των δικαστών, αρχές του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε επίσημη γνωμοδότηση, υποστήριξε απόλυτα την πρόταση του δικαστηρίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή τη φορά δεν είναι αυτή που κάνει την πρόταση, αλλά είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου. Και ε, την αφορά άμεσα, διότι μεγάλος αριθμός των αποφάσεων αυτών, ε, διαφόρων αποφάσεων, αμφισβητούνται από, και βρίσκουν απάντηση στο δικαστήριο. Δεν είναι η μόνη που υποστήριξε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θυμόσαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξίσου υποστήριζαν αυτή την πρόταση για την αύξηση του αριθμού των δικαστών και μόνο οι δυσκολίες που αφορούσαν την επιλογή των ε, προσδιορισμών ε, δικαστών εμπόδισε την υλοποίηση της πρότασης. Εν τω μεταξύ, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου, αυξήθηκε ο αριθμός των υποθέσεων στο δικαστήριο, αυξήθηκε σημαντικά και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως το δικαστήριο και φρονεί ότι οι νέες ιδέες που παρουσιάστηκαν από αυτό ε, είναι καλές. Αρκούν για την κάλυψη του προβλήματος. Κυρίως διότι η πρόταση του δικαστηρίου είναι απρόταση που δίνει σταδιακή απάντηση ανάλογα με την τάση των εκδικαζομένων υποθέσεων. Προβλέπονται τρία στάδια, ολοκληρώνεται η δικασία το 2019. Σταδιακά λοιπόν λέγω το δικαστήριο θα αυξήσει το δυναμικό του. Ε, εν συντομία να προσθέσω δύο στοιχεία, αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ίσως το μόνο σημείο επί το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε παρατήρηση ή κάποιες κρίσεις εξέφρασε όσον αφορά την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και συμπεριλαμβάνεται στην γνωμοδότηση του 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλωστε αυτή η άποψη που αναφέρω. Πιστεύει ότι ένα δικαστήριο κυρίως σε ένα δικαστήριο με 56 δικαστές θα πρέπει να αλλάξει ριζικά τις μεθόδους εργασίας του. Και πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η βασική αρχή που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το δικαστήριο είναι η αρχή της εξειδίκευσης ε, όσον αφορά τις αποφάσεις. Βλέποντας το τεχνικό χαρακτήρα, τον περίπλοκο χαρακτήρα των υποθέσεων, θα πρέπει το δικαστήριο να διοργανωθεί ε, τα διάφορα σχήματα του δικαστηρίου κατά ειδικότητα. Και η κάθε ειδικότητα του δικαστηρίου, του κάθε τμήματος δικαστηρίου να ασχολείται με τις διάφορες συγκεκριμένες υποθέσεις. Και το δεύτερο, άκουσα να αναφέρεται η εναλλακτική ιδέα που συζητείται καμιά φορά. Δηλαδή, το δικαστήριο δεν χρειάζεται παραπάνω δικαστές, αρκεί να αυξηθούν οι συνεργάτες των δικαστών. Αν επιτρέπεται μία αντίδραση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά κάποιον που ασχολιόταν με τις παραπομπές υποθέσεων στο δικαστήριο, οι δικαστές του ε, δικαστηρίου πολύ συχνά αντιμετωπίζουν κάθε εβδομάδα δύο-τρεις ημέρες ακρόασης. Ολόκληρη ημέρα συζητήσεων μεταξύ δικαστών για να ετοιμάσουν τις αποφάσεις και ο χρόνος που απομένει σε κάθε δικαστή θα πρέπει να αφιερώνεται στην, απο... στην εξέταση σχεδίων αποφάσεων. Έχει τι συνεργάτες ο κάθε δικαστής. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάζει και να επεξεργάζεται κάθε δικαστής το έργο τριών συνεργαστών συνεργατών, συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα επιμακρών υπάρχουν αυτοί οι τρεις συνεργάτες στο δικαστήριο. Ο φόρτος εργασίας σε κάθε δικαστή ε, δεν το επιτρέπει ε, να είναι μεγάλος αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πάνω από ε, τρεις βοηθούς. Άμα έχει πέντε βοηθούς δεν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά επανεξέτασης των διαφορών προτάσεων που τυποβάλλονται. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε νομίζω το αντικείμενο. Η νέα διαπραγματευτική ομάδα συμφωνήθηκε ότι πέραν της διαπραγματευτικής εντολής που εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2013 η διαπραγματευτική ομάδα συντίθεται ως εξής επικεφαλής Σόβοντα με μέλη Ντεπίντου και Σφιεύκα και κυρία Χαουτάλα. Αυτά σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση που και Θα έρθω στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, που είναι το υπαριθμό 35. Και θα ήθελα, μια και δεν βλέπω τον κύριο Καβαδά, εδώ να δώσω τον λόγο στον κύριο Τσαμπάσκι. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω όμως βουλγαρικά. αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο ευρωπαϊκή Διακόπτη, με συγχωρείτε, φαίνεται προϋποθέσεις υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζουμε ότι οι συναδελφοί μας δεν είχαν πατήσει τόσο στο κουμπί. Έχει καλώς. Ας αρχίσουμε λοιπόν και πάλι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έλεγα πριν, είχα την τιμή να είμαι παρόν στην ετήσια συνέλευση για θέματα διανοητικών δικαιωμάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων στο Αλικάντε της Ισπανίας το Νοέμβριο που μας πέ... φέτος μάλλον και μαζί μου ήταν και ο κυρίος Καβαντά η παρουσία μας εκεί αποδείχθηκε σημαντική διότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να είναι παρόν ως παρατηρητής και οι ευρωβουλευτές μάλιστα είναι καλόδεκτικοί ως εκπρόσωποι Και άλλωστε είμαστε σημαντικοί εκεί και για τον ιδιωτικό τομέα και για τον δημόσιο. Πάντως η επίσκεψή μου ήταν χρήσιμη, συνέλεξα πολλές πληροφορίες. Το παρατηρητήριο ιδρύθηκε το 2009 με στόχο να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την παραποίηση διαφόρων προϊόντων, πώς αυτή η παραποίηση, η πλαστογράφηση κλπ ε, επηρεάζουν την οικονομία και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν. Η Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο εισηγητής της κ. Μάση Ντάλγο των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κατέληξε σε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του παρατηρητηρίου διανοητικών δικαιωμάτων και έτσι αναλαμβάνει νέα καθήκοντα το γραφείο σημάτων του Αλικάντε. Ένα από τα στοιχεία στα οποία κατέληξαν στις διαπραγματεύσεις αυτές ήταν η αλλαγή του τίτλου του παρατηρητηρίου. Λεγόταν Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Πειρατεία και Παραποίηση και τώρα λέγεται για την παραβίαση δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή διανοητικών δικαιωμάτων. Εμείς ε, λάβαμε υπόψη και πληροφορίες που έχουν σχέση με κάποιες μελέτες και ε, από αυτές τις πληροφορίες θα σας πράγματα. Από τον Οκτώβριο του 2012 που άρχισε το έργο του παρατηρητηρίου έχουν ε, εκτελεστεί σημαντικά πράγματα. Έχουν συλλεχθεί πολλά σημαντικά στοιχεία προς πληροφόρηση μας μόνοι δηλαδή που λαμβάνουμε τις αποφάσεις, αλλά και για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. και για να διευκολυνθεί το έργο των κυρίων των ε, διανοητικών δικαιωμάτων. Είναι διάφορες μελέτες Πρώτα για τους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι από την άποψη αυτή, επίσης πώς επηρεάζεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μία από τρεις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται άμεσα με την προστασία των ειδικών δικαιωμάτων. το, η απόδοση του τομέα αυτού ανέρχεται στο 39% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως απασχολούνται στο τομέα αυτό μικρές και μεσές επιχειρήσεις, οι οποίες εποφελούνται κιόλας από την προστασία των ε, δικαιωμάτων βιομηχανικής διοκτησίας αντίθετα από την κυριαρχούσα άποψη που θεωρεί ότι ε, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις εποφελούνται από αυτό. Διερευνήθηκαν επίσης και οι απώλειες, οι ζημίες δηλαδή, από την παραποίηση κυρίως καλλιντικών, που αυτές ανέρχονται σε 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και θίγονται 50.000 θέσεις απασχόλησης. Άλλη μελέτη εξέτασε το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες την βιομηχανική διοκτησία ή τα διανοητικά δικαιώματα. Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι είναι σημαντικά τα πράγματα αυτά και η συνειφορά τους στην οικονομία. Όμως όταν μιλούν για τις προσωπικές τους συνήθειες και την προσωπική τους στάση, πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι ε, κάποιες μικρές παραβιάσεις δικαιωμάτων ε, πνευματικών ε, δικαιωμάτων, ε, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είναι δικαιολογημένη, γιατί είναι, δύσκολο, είναι ακριβό το να κατεβάζει κανείς πράγματα από το ίντερνετ νομίμως και ούτω καθεξής. Και όλων ότι τελικά δεν υπάρχει και μεγάλο κακό να το κάνουν. Αυτές οι απόψεις μάλιστα είναι ευρύτατα διαδεδομένες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών 15 έως 24 ετών. Επίσης, οι τράπεζες δεδομένων επιβολής, enforcement database, χρησιμοποιείται πολύ από τους κατόχους των ε, δικαιωμάτων και υπάρχει και μετάφραση. Η βάση δεδομένων άρχισε να λειτουργεί από τα τέλη του 2013 και χρησιμοποιείται ήδη ευρύτατα. Είναι μάλιστα προσβάσιμη και σε τελωνιακές αρχές. Είναι σημαντικό εργαλείο και διευκολύνει πολύ τους κατόχους των δικαιωμάτων να εξασφαλίσουν σεβασμό των δικαιωμάτων τους και να έχουν και καλύτερη πρόσβαση στους οργανισμούς επιβολής του δικαίου. Υπάρχουν όμως και έργα τα οποία βρίσκονται σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες κλπ. των οποίων οι δημιουργοί δεν μπορούν να βρεθούν. Το ίδιο ισχύει και για ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Υπάρχει θετική οδηγία, η 28-2012, που προβλέπει τη δημιουργία ενός ενίου μητρώου όλων των ανοιχτών έργων πανευρωπαϊκού. Και κάθε έργο που θα περιλαμβάνεται εκεί θα μπορεί να χρησιμοποιείται από πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικούς φορείς, με εξασφάλιση ταυτόχρονα των δικαιωμάτων. Αυτή η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί από το ίδιο το παρατηρητήριο σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους Υπάρχει λοιπόν αυτή η βάση δεδομένων, έχει αρχίσει να λειτουργεί από τον Οκτώβριο και οι δημιουργοί της μου την παρουσίασαν με αρκετή υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν οι εντυπωσει μου αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι από την επίσκεψη αυτή είναι ότι το παρατηρητήριο είναι σημαντικό, πολύ χρήσιμο και να παρακολουθούμε το έργο του να χρησιμοποιούμε τα συμπεράσματα των εργασιών του παρατηρητηρίου για το έργο μας. Και για το λόγο αυτό προσκάλεσα μάλιστα τον ίδιο τον πρόεδρο Καμπίνος, βεβαίως την πρόσκληση αυτή πρέπει να τη συζητήσουμε και εδώ, να προσέλθει σε συνάντηση της Επιτροπής μας και να μιλήσει για το έργο του παρατηρητηρίου του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχουν κάποια σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής. Δεν φαίνεται. Θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεμάσκης. Περνάμε στο σημείο 36 και η κυρία Χαούταλα ο συζήτης έχει έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μην είμαι εξαρτητική, αντίθετα να είμαι σύντομη και συνεκτική. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω οκτώ σχέδια εκθέσεων που έχουν ταυτόσιμο χαρακτήρα και έχουν να κάνουν με την προσχώρηση οκτώ κρατών στην σύμβαση της Χάγης του 1998 σε ό,τι αφορά τις ε, αστικές πτυχές της ε, απαγωγής τέχνων η λεγόμενη σύμβαση της Χάγης. Τα περισσότερα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια μετά από τις αιτήσει γονέων των οποίων τα παιδιά έχουν απαχθεί και έχουν πάει σε τρίτες χώρες. Τα υψηλά συμβαλόμενα ε, μέλη τώρα είναι η Ανδόρα, η Αλβανία, η Γκαμπόν, Ρωσία, Σεϊχέλες και η Σιγκαπούρη. Οι χώρες αυτές θέλουν τώρα λοιπόν να προσυπογράψουν αυτή τη σύμβαση ως συμβαλόμενα μέλη. Φυσικά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κυρώσει αυτή τη σύμβαση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει καθυστερήσει η προσχώρηση των χωρών αυτών το 2011 λόγω νομικών αβεβαιοτήτων που έχουν καθυστερήσει την ε, είσοδο αυτών των νέων κρατών. Δεν ήταν σαφές το αν η αποδοχή αυτών των κρατών ήταν της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ου. Η Κομισιόν έδωσε μια πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με την αποδοχή αυτών των χωρών ήδη το Δεκέμβριο του 2011. Το Συμβούλιο όμως δεν ενέκρινε αυτές τις προτάσεις λόγω της αμφισημίας σε σχέση με το θέμα της αρμοδιότητας. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν υποστηρίξει την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, ενώ κάποια κράτη στο Συμβούλιο δεν συμφώνησαν. Το 2013 το θέμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεπέμφθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για γνωμοδότηση και πριν από ένα μήνα το δικαστήριο έδωσε μια απάντηση. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στα εξωτερικά θέματα για τον τομέα αυτό, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι η σύμβαση αυτή δεν επιτρέπει την αυτόνομη δράση διεθνών οργανισμών. Λοιπόν, χρειάζεται μια απόφαση του Συμβουλίου, επομένω, η οποία ζητά από τα κράτη-μέλη να αποδεχθούν την προσχώρηση νέων συμβαλωμένων μερών στη Σύμβαση της Χάγης. Εν συντομία τώρα θέλω να σας παρουσιάσω τα κύρια στοιχεία αυτής της σύμβασης. Εισάγει τον λεγόμενο μηχανισμό επιστροφής και αυξάνει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Ο μηχανισμός επιστροφής είναι μια διαδικασία που έχει αποφασιστεί για να εξασφαλιστεί η ταχεία επιστροφή των απαχθέντων παιδιών στην χώρα και την αιστεία τους. Προβλέπει η Σύμβαση επίσης μέτρα διοικητικής συνεργασίας για να μπορέσει να διακριβωθεί η ταυτότητα και η προέλευση των παιδιών και εξασφαλίζει ότι οι νόμοι οι οποίοι θα εφαρμοστούν αυτή της χώρας διαμονής του παιδιού. Επίσης προωθεί την δυνατότητα επαφών ώστε το παιδί να μπορέσει να διατηρήσει επαφέ με τον γονέα ο οποίος μένει έξω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά η Σύμβαση ήταν επιτυχής και έχει συμβάλει τα μάλα στο να επιληθούν πολλέ υποθέσει απαγωγή παιδιών. Πρέπει να χαιρετήσουμε λοιπόν ιδιαίτερα την προσχώρηση των νέων συμβαλωμένων μερών τώρα που έχει αρθεί η αμφισημία σε σχέση με την νομική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό, με την προσχώρηση αυτή έχουμε καλύτερες διασφαλίσεις εναντίον των απαγωγών παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν απαχθεί στις 8 αυτές χώρες Αρμενία, Ανδόρα, ε, Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες διμερείς συμφωνίες για ορισμένα κράτη-μέλη και λόγω αυτής της καθυστέρησης πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με τις νέες συμβαλόμενες χώρες ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ήδη τις ρήτρες της σύμβασης ενώ εκρεμεί η Ευρωπαϊκή ε, ρύθμιση του θέματος αυτού. Η Φιλανδία, παραδείγματος χάρη, έχει εφαρμόσει αυτή τη σύμβαση με τη Ρωσία ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013 από τη βάση μιας διμερούς συμφωνίας με τη Ρωσία. Εν κατακλείδη λοιπόν ως εισηγήτρια για τα θέματα αυτά υποστηρίζω απόλυτα την προσχώρηση αυτών των νέων κρατών και προτείνω το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τις προτάσεις αυτές ώστε να υπάρξει η απόφαση του Συμβουλίου για κάθε μία από αυτές τις χώρες. Αλλά, αλλά υπήρξε μία δυσάρεστη καθυστέρηση στη διαδικασία από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι η άποψη της νομικής υπηρεσίας, αν υπάρχουν κάποια ε, νομικά μέτρα που μπορούν να λυθούν για να μειωθεί αυτή η καθυστέρηση. Επιτρέπει η Σύμβαση μια αναδρομική εφαρμογή των ε, προνοιών αυτής σε περιπτώσεις απαγωγής παιδιών που έχουν γίνει μεταξύ του 2012 και του 2014 θα ήταν πολύ σημαντικό για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Σχόλια. Κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Η νομική υπηρεσία έχει απάντηση για την ερώτηση της ε, κυρίας Χαουταλα. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα και για την ώρα η νομική υπηρεσία δεν έχει απάντηση. Βεβαίω μπορούμε να μελετήσουμε το θέμα και να επανέλθουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης εσάς κυρία Χαουτάλα και ας περάσουμε τότε στο τελευταίο θέμα του σημερινού πρωινού που είναι το υπαριθμό 37 σχετικά με την επικουρικότητα. και δύο αιτιολογημένες γνώμες από δύο εθνικά κοινοβούλια, των οποίων ήταν το κρατικό, το άλλο δεν το ακούσαμε. Δεν έχουμε την διαρκή εισηγήτρια κυρία Ντελβό κοντά μας, αλλά της έχει ζητηθεί η γνώμη και δεν έχει να υποβάλει κανένα σχόλιο σχετικά με αυτές τις αιτιολογημένες γνώμες. Αν και από εσά μέλη δεν υπάρχουν σχόλια. Αυτό σημαίνει τότε ότι ολοκληρώσαμε για σήμερα το πρωί. Σας εύχομαι καλή όρεξη και θα τα πούμε στις 3.